Καθίστε παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας μετά τις διακοπές. Πρώτα τα τυπικά, έγκριση δηλαδή της ημερήσιας διάταξης, οι ανακοινώσεις της Προέδρου θα γίνουν μετά τον κύριο Ντάισελ Οπότε θεωρώ ότι εγκρίνεται την ημερήσια διάταξη και σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε εγκρίνει και τα πρακτικά της συνεδρίασης 8-9 Ιουλίου 2013. Θεωρώ ότι έχουν ε, εγκριθεί γιατί έχουν διανεμηθεί όσοι ήθιστε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα προχωρούμε στην ακρόαση με τον πρόεδρο της Ευρωομάδας. Αυτό είναι μέρος μια σειρά ανταλλαγών στα πλαίσια του οικονομικού διαλόγου και θυμίζω στα μέλη ότι εστιάζομαι σε συστάσεις συγκεκριμένες για χώρες στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ιδιαίτερα ε, πρέπει να συζητήσω με δημοσιονομικές ε, και μακροοικονομικές ε, προκλήσεις, δυσκολίες και συστάσεις στα πλαίσια του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2013 που ενέκρινε τον Ιούλιο το Συμβούλιο. Και θα μας πει ο Υπουργός για όλα αυτά. Είναι η τρίτη επίσκεψη στην Επιτροπή μας ε, του κυρίου Ντάισελμπλουμ. Ε, είχαμε δύο τακτικούς οικονομικούς διαλόγους και σύν την πρόσθετη επίσκεψη για την Κύπρο. Καλώς ήρθατε, σας αισθανόμαστε πια σαν παλιό φίλο και σας δίνω το λόγο για να μας κάνετε τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις για τις συστάσεις που είναι ειδικέ για κάθε χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να έχω μαζί σας για μια ακόμη φορά με ανταλλαγή απόψεων με θέμα αυτή τη φορά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τις συστάσεις αναχώρα συνολικά για την Ευρωζώνη. Στην πρώτη μου παρουσία ενώπιον τη επιτροπή σα είχα πει ότι είμαι φιλόδοξο. Θέλω από την διαχείριση της κρίσης να περάσουμε ε, σε μια πιο θεμελιώδη προσέγγιση, δομική προσέγγιση για την ενίσχυση της οικονομίας, της λειτουργία ε, της οικονομίας της Ευρωζώνης. Και βέβαια, ξακολουθεί να είναι μακρύ ο δρόμο που έχουμε να διανύσουμε. Χαίρομαι όμω γιατί βλέπω ότι το μονοπάτι που ακολουθούμε μα φέρνει μακριά από την κρίση σε μια πολύ αναγκαία δομική συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τι συστάσει αναχώρα, τι είδαμε πριν το καλοκαίρι στο Eurogroup. Ομόφωνα δε τα κράτη-μέλη της ενέκριναν και είναι σημαντικές, ε, ε, οι, μάλλον οι σημαντικοί τομείς ε, επισημάνθηκαν κάποιου από του οποίου θα σας αναφέρω, κάποιε από τις συστάσεις συγκεκριμένα. Πρώτη σύσταση είναι η ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου που ισχύει για τα μέλη της Ευρωζώνης. Επίσης θέλουμε να υπάρχει παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων για να είναι συνεκτική η οικονομική πολιτική. Δεύτερη σύσταση, παρακολούθηση, συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής ε, των κρατών μελών της Ευρωζώνης ε, για να έχουμε διαφορετικές ε, δημοσιονομικές πολιτικές που είναι όμως φιλικές προς την ανάπτυξη. Τρίτον, να δούμε γιατί είναι διαφορετικά τα επιτόκια δανεισμού, ιδίως προς τις ΜΜΕ και να δούμε ο κατακαιρματισμός των αγορών πώς μπορεί να καταπολεμηθεί για να ξεπεράσουμε τις αρνητικές τάσεις. Τέταρτη σύσταση, ήταν ε, η ισοσκέληση του υπολογισμού. Θέλαμε ε, οι τράπεζες ε, να καταφέρουν να βελτιώσουν τους ισολογισμούς τους και να μην έχουμε κατακαιρματισμό, να, έχουμε να επανέλθει η κανονικότητα και η ομαλότητα στο δανεισμό. Πέμπτη σύσταση είναι τα μεταρρυθμιστικά σχέδια, τα, τα σχέδια για μείζονες μεταρρυθμίσεις. Είπαμε ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στο συντονισμό του εξάντε, του εκπροντένου συντονισμού των ε, μεγάλων οικονομικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη. Και η τελευταία έκτη ε, σύσταση ήταν να αντιμετωπιστούν και οι τελικές επιπτώσεις της κρίσης, ιδίως ό,τι αφορά την ανεργία των νέων. Αυτές οι συστάσεις συνάδουν απόλυτα με τις προτεραιότητες του Eurogroup και νομίζω ότι έχουμε ήδη ε, τα βασικά στοιχεία, τα βασικά δομικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Με το Six Pack έχουμε καλύτερο συντονισμό, καλύτερη εποπτεία στην οικονομική και δημοσιονομική πολιτική όλων των κρατών μελών Κάτι που είναι ιδίω σημαντικό για την ε, Ευρωζώνη είναι οι διαδικασίες μακροοικονομικών ανισορροπιών. Εμείς παρακολουθούμε το μηχανισμό ελέγχου ε, και ειδοποίησης ε, και συναγερμού της Κομισιόν, ε, όπου εντοπίζονται ανισορροπίες, τις παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Θέλουμε να εντοπίσουμε τις ανισορροπίες, εκεί που είναι υπερβολικές, οι μακροοικονομικές αυτές ανισορροπίες, μια διαδικασία που δείχνει ότι χρειάζεται ακόμη προσαρμογή στις οικονομίες μας. Πρέπει να διατηρηθεί η όθηση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και στην αγορά προϊόντων. Το Tupac τώρα ε, άρχισε να ισχύει αφού είχαν εκπονηθεί οι συστάσεις που σας προανέφερα και θα είναι πάρα πολύ σημαντική νομοθεσία αυτή για το συντονισμό ε, του οικονομικού και δημοσιονομικού προγραμματισμού στα κράτη-μέλη. Γίνονται τώρα τα απαραίτητα ε, σχέδια, έχουμε έτσι ε, ανεξάρτητες προβλέψεις και στα κράτη-μέλη. Όλα αυτά θα τα μελετήσει πάρα πολύ προσεκτικά η Κομισιόν μεμονωμένα για κάθε χώρα και με βάση τις αναχώρας συστάσεις. Επίσης και το, τη διαδικασία ε, περιβολικού ελλείμματος, το σύμφωνο ε, ανάπτυξης, βλέπουμε τους στόχους και αν δούμε να μην υπάρχει ε, συμμόρφωση και αυτό να διαρκεί, τότε το εν λόγω κράτος μέλος ενδεχομένως θα κληθεί να υποβάλει ένα αναθεωρημένο σχέδιο για αυτό το φθινόπωρο. Σε ό,τι αφορά τώρα τι απόψει Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο προπολογισμού και για τι επιπτώσει που θα έχει για την Ευρωζώνη, ε, θέλω λοιπόν να του δώσω πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο Eurogroup. Θα τα συζητήσω όλα αυτά με του υπουργού σε μια συνεδρίαση τη Eurogroup που θα είναι αφιερωμένο σε αυτό το θέμα και θα λάβει χώρα το Νοέμβριο. Οι απόψει ε, επομένω ε, του Eurogroup θα ληφθούν υπόψη, ελπίζουμε, πριν ε, την κατάρτιση των εθνικών προπολογισμών στα τέλη της χρονιάς. Τώρα, διευκόλυνση δανεισμού των επιχειρήσεων για να μπορούν να κάνουν παραγωγικέ επενδύσει, να παραμείνουν παραγωγικέ. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα σχεδόν σε όλε τι χώρε μα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Νομίζω ότι είναι γνωστό τη σπάση ότι οι ΜΜΕ είναι κεντρικές, είναι πολύ σημαντικές για την ανάκτηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων μετά την αύξηση κεφαλαίου την άνοιξη έχει ρόλο σημαντικό να διαδραματίσει και ελπίζουμε να δώσει μεγαλύτερη στήριξη στις ΜΜΕ σε όλη την Ένωση. Επίσης το Μάιο συστάθηκε μια ομάδα ε, ε, εμπειρογνωμών υψηλού επίπεδου που θα βλέπει τη ε, χρηματοδότηση των ΜΜΕ και περιμένουμε και τι συστάσει αυτής τη ομάδας. Νομίζω θα είναι και στο ECOFIN, στην μέση σχεδιάτηση του ECOFIN στο Βίλνιους το θέμα αυτό. Πρόσφατα άλλα μέτρα, οι βήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ασθενή συνεργασία με την Κομισιόν, και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν να συζητήσουμε πώς χρηματοδότηση, η τραπεζική χρηματοδότηση προς τις ε, ΜΜΕ μπορεί να βελτιωθεί. Ε, θα κορυφωθούν με μια έκθεση που θα ε, υποβληθεί το Σεπτέμβριο στο ΕΚΟΦΗΝ σχετικά. Είναι πρωτοβουλίες όλες αυτές που θα συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Ουσιαστικά θέλουμε να ολοκληρώσουμε όμως την Τραπεζική Ένωση, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ε, μακροχρόνια σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, θα πάψει ο κατακαιρματισμός και θα επανέλθει ε, στα κανονικά του, στα ομαλά επίπεδα η διαδικασία δανεισμού και προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε όλα τα θέματα για την Τραπεζική Ένωση, το Single Rule Book, ε, η βελτίωση της εποπτείας. Ε, είναι θέματα που δεν μπορούν να περιμένουν. Ε, είχαμε ένα θετικό βήμα πρόσφατα που ήταν η έγκριση της τέταρτης οδηγίας για τις κεφαλικές απαιτήσεις, το CDR4. Έχουμε επιτυχίες, πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτές και θα προσπαθήσουμε και εμείς να οργανώσουμε όλες τις διαδικασίες ώστε και η οδηγία για το BRD, ε, για το Ταμείο για την Καθάριση των Τραπεζών να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Ε, στόχος είναι να προστατεύσουμε το φορολογούμενο από πάρα πολύ δαπανερά σχέδια διάσωσης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο το ποιοι θα συμμετέχουν σε μια διαδικασία καθάρισης ή διάσωσης τράπεζας και σε ποιο βαθμό καθένας. Αυτός ε, ο μηχανισμός, ο νέος εποπτικός μηχανισμός είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει να λειτουργεί από του χρόνου. Ε, την, ε, τις μεγάλες τράπεζες ένωσης θα τις επιβλέπει από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ενίο εγχειρίδιο κανόν, το Single Rule Book, θα αρχίσει να ισχύει σύντομα παντού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη ε, να έχουμε μια νέα αντιμετώπιση και στα διασυνοριακά ζητήματα. Και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα προβεί σε μια αξιολόγηση των τραπεζών πριν αρχίσει να ισχύει ο ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και αν εκεί ανοιχνευθούν προβλήματα για κάποια τράπεζα, θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για το ποιος θα απομειστεί ε, την ευθύνη ε, και το κόστος ε, για τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Έχουμε και το μέσο για την άμεση ανακεφαλοποίηση. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το, αυτή η νομοθεσία. αλλά μπορεί να ισχύσει αυτή η άμεση ανακεφαλοποίηση πριν έχουμε αυτόν τον ενιαίο μηχανισμό για την ε, καθάριση των ε, τραπεζών. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε. Και χαιρετίζω το γεγονός ότι τώρα έχουμε συγκεκριμένη πρόταση για να συζητήσουμε ε, αυτό το θέμα, να έχουμε και ένα ενιαίο ταμείο και ένα ενιαίο συμβούλιο για την εξυγίανση ε, των ε, τραπεζών. Ο στόχος μας είναι σαφής και δεν πρέπει να ε, ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό για την εξυγίανση των τραπεζών που έχουν αποτύχει. Για να μειωθούν δε, για να μειωθεί δε το κόστος πρέπει και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Και φυσικά ο απότερος στόχος είναι η προστασία των φορολογουμένων. Members, πριν απαντήσω στις ε, ερωτήσεις σας, ε, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το ελληνικό πρόγραμμα που συζητάτε εντατικά. Ιδίως στη διάρκεια του καλοκαιριού συζητήθηκε πάρα πολύ. Όπως βλέπω την κατάσταση είναι η Εξή, τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος έγινε τον Ιούλιο με αποτέλεσμα να ε, δούμε ότι είναι στο σωστό δρόμο, βελτιώνεται η κατάσταση η ελληνική οικονομία θα γυρίσει σε επίπεδα ανάπτυξη μάλλον στι αρχέ τη επόμενη χρονιά και οι ελληνικέ αρχέ σημειώνουν σημαντική πρόοδο υπό πολύ δύσκολε συνθήκε για την ε, οικονομική βιωσιμότητα, για την υλοποίηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα τη οικονομία. Όμω απαιτείται περαιτέρω πρόοδο, ιδίω στον τομέα ε, των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα και ε, στον τομέα τη διαχείριση τη φορολογία. Η δεύτερη αναθεώρηση θα γίνει φέτο και όταν ολοκληρωθεί θα έχουμε μια επικαιροποιημένη έποψη για την υλοποίηση του προγράμματος και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του τρέχοντος προγράμματος. Και αυτό το θέμα θα μπει στην ημερήσια διάταξη ε, τον επόμενο μήνα και αυτή η διαδικασία θα, ε, το, το σκέλος αυτής της διαδικασίας θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ενδεχόμενο να χρειαστεί νέο τρίτο πρόγραμμα, ε, τρίτο μνημόνιο, παρά την πρόοδο είναι σαφές ότι τα προβλήματα της Ελλάδας δεν έχουν εντελώς ή δεν θα έχουν εντελώς επιληθεί μέχρι το 2014. Επομένως είναι ρεαλιστικό να σκεφτούμε ότι θα χρειαστεί περαιτέρω στήριξη πέραν αυτού του προγράμματος. Σε αυτά τα πλαίσια το Eurogroup ξεκάθαρα δήλωσε ότι δεσμεύεται να παράσχει την αναγκαία επαρκή υποστήριξη στην Ελλάδα και στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού μέχρι να ξαναγυρίσει στις αγορές η Ελλάδα. Βέβαια θα πρέπει η Ελλάδα να ε, εφαρμόσει πλήρως όρους του προγράμματος και ε, το 2014 θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το κατά πόσο εφαρμόζονται πλήρως όλοι οι ε, υπήρξε πολλή οικοτολογία και εικασίες και συζητήσεις ε, ε, στα μίντια για το κατά πόσο θα μπορούσαν να μειωθούν ε, τα επιτόκια ε, στο μέσο ε, για τη διευκόλυνση δανεισμού ή η χρηματοδότηση εδρετικών ταμείων. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να πληρούνται και κάποιοι όροι. Δηλαδή, αν μπορούμε να έχουμε μία μείωση κάποιων επιτοκίων και όρων δανεισμού. Πάντως ε, δεν μπορούμε να εξελίσσουμε τα πόσον αυτές οι συνθήκες ε, πληρούνται προς κάτι τέτοιο. Αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε τον Απρίλιο του 2014 και όλα αυτά τα είχαμε συμφωνήσει το Δεκέμβριο. Τον Απρίλιο, τον νωρίτερο λοιπόν, θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την πρόοδο του μνημονίου του προγράμματος και να δούμε κατά πόσον ε, υπάρχει βιωσιμότητα του χρέους. Και γι' αυτό δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή να κάνουμε εικασίες Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι έτοιμος να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρουσιάσατε έτσι ευρέως κάποια θέματα. Ελπίζω να μπορέσουμε να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα το SSM στη, τον ενιαίο αποπτικό μηχανισμό στο Στρασβούργο. Περιμένουμε το τελικό κείμενο από την ΕΚΤ για την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά έγινε πρόοδος σε αυτό το μέτωπο και συνεχίζονται οι τριμερείς διάλογοι για την οδηγία διάσωσης και εξυγίανσης των τραπεζών, και θα παρουσιάσουμε τα θέματα αυτά αργότερα. Τώρα, ένα σημαντικό κομμάτι του SSM, του ενιαίου Ποπτικού μηχανισμού, είναι η εξέταση από την ΕΚΤ της ποιότητας των ε, στοιχείων του ενεργητικού. Υπάρχουν κάποιες πιέσεις, σύμφωνα με φήμες, σχετικά με τη συμμετοχή του πρωτογενού στο ΜΕΑ ε, ή ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και ενεργό συμμετοχή του. Αυτό προέρχεται από κάποια, κάποιους τομείς. Και δεν ξέρω, έχετε εσείς κάποια ιδέα, συζητείτε το θέμα στην Ευρωομάδα ή έχετε προσωπική άποψη. Νομίζω ότι η άποψη δική μου και των μελών είναι ότι η διεθνής σκηνή περιμένει να υπάρχει μία σε βάθος και πολύ δραστήρια συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ούτως ώστε να υπάρχουν ξεκάθαρα τα πράγματα, να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τα κληροδοτούμενα και να ε, κάνουμε ένα πρώτο βήμα προς την επιτυχία. Βεβαίως αυτό δεν ε, υπονοεί κάτι κατά της ΕΚΤ. Απλώς είναι η προσδοκία των διεθνών αγορών. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το σχολιάσετε και αυτό το πρόσθετο στοιχείο που σας έδωσα πριν πάμε στην ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γίνει σωστή αρχή με την Τραπεζική Ένωση και η πρώτη αρχή θα είναι του χρόνου το φθινόπωρο όταν αρχίσει την εποπτική της δραστηριότητα στις μεγάλες τράπεζες, η Κεντρική Τράπεζα. Θέλω με πλήρη αξιολόγηση των ισολογισμών που αποτελείται από δύο μέρη. Ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων και το stress test από την Τραπεζική Αρχή και την ΕΚΤ. Αντίστοιχα, να ξεκαθαρίσω ότι πρέπει να είναι διεξοδικός ο έλεγχος και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για την ποιότητα του ελέγχου αξιολόγησης και είναι σημαντικό από, και για πρακτικούς λόγους ε, ότι σε ένα χρόνο πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και χρειάζεται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Οπότε και από πρακτικής πλευράς θα ήταν σημαντικό να έχουμε τη συμμετοχή τους. Δεν ε, το συζητήσαμε στην Ευρωομάδα αυτό. Δεν νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθεί η αξιολόγηση των ισολογισμών θα είναι θέμα πολιτικών πιέσεων ή αντικείμενο πολιτικής συζήτησης, θα γίνει ανεξάρτητα, ε, διεξοδικά και δεν τίθεται θέμα για την ποιότητα της δουλειάς που πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει όμως καλή αρχή με την Τραπεζική Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ε, καλά αυτά που μας λέτε, μας διαβεβαιώνουν για την καλή πορεία του πράγματος. Ε, φαντάζομαι και οι συνάδελφοι θα συμφωνούν. Υπάρχουν και νέα μέλη που θα συμμετέχουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Υπενθυμίζω τους κανόνες. Πέντε λεπτά θα ε, έχετε για να κάνετε τις ερωτήσεις σας και πέντε λεπτά για την απάντηση. Αν ξεπεράσετε το χρόνο σας δεν θα πάρετε απάντηση. Αν ε, μιλήσετε σύντομα θα μπορείτε να ξαναλάβετε το λόγο για να προσθέσετε κάτι σε μισό λεπτό. Ε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Εμείς ε, ε, νομίζω θα τα καταφέρνουμε καλά. Από την κυρία Βόρτμαν Κόλ από το ΕΛΚ η πρώτη ερώτηση. Ως εισηγήτρια του Six θέλω να σας ε, ευχαριστήσω για την ευθύνη που αναλάβατε και την υπευθυνότητα για την εφαρμογή των συστάσεων για κάθε χώρα. Οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικές για την οικονομική ανάκαμψη και την απασχόληση. Και μπαίνουμε το φθινόπωρο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση όπου η Κομισιόν θα αξιολογήσει τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και του Ολλανδικού προϋπολογισμού και είναι καλό που μας λέτε ότι στην Ευρωομάδα ε, δραστήρια λαμβάνετε υπόψη τι συστάσει για τον προπολογισμό. Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων είναι σημαντική. Η ερώτησή μου αφορά την Τραπεζική Ένωση όμω. Φέτο, πριν αρχίσει η εποπτεία από την ΕΚΤ, μιλήσατε ήδη για τον έλεγχο τη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, των στοιχείων του ενεργητικού, που δεν θα είναι πολιτικό θέμα, αλλά πώ θα διασφαλίσετε ότι ο έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων θα είναι ανεξάρτητο γιατί αυτό είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε την ανεξαρτησία του ελέγχου. Και τι θα γίνει αν ας πούμε υπολείπεται μια τράπεζα, αν δεν τα καταφέρει, αν δεν είναι εντάξει. Υπάρχει σχέδιο άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αλλά πότε θα γίνεται αυτή. Και πώς θα χρησιμοποιείτε, γιατί πάντα λέγατε ότι θα πρέπει να πληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό και πώς θα χρησιμοποιείται ο ESM σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ θέλω να υπάρχει αυτή η προστασία, αυτό το backstop, αλλά πώς θα γίνεται. Και τελευταία ερώτηση αφορά τον ενιαίο μηχανισμό εκαθάρισης. Ε, χαίρομαι που στηρίζετε την πρόταση της Κομισιόν γιατί έτσι ερμήνευσα τα σχόλια που μας κάνατε μόλις τώρα. Αλλά ο κόσμος ε, και τα ΜΜΕ, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, λένε ότι κάποιοι σημαντικοί υπουργοί οικονομικών είναι κατά του ενιαίου κομματιού του SRM. Αλλά να είναι ενιαίος ο μηχανισμό ε, είναι πολύ σημαντικό, όπω είπε και ο πρόεδρο Δράγκη, είναι σημαντικό πυλώνας στα πλαίσια τη Τραπεζική Ένωση. Αυτό πώ θα το χειριστείτε και πιστεύετε ότι θα περάσει η πρόταση τη Κομισιόν από την Ευρωομάδα και του Υπουργού Εκοφήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ε, τις ερωτήσεις σας, ε, κυρία Βόρτμαν Κόλ. Όχι, θα μιλήσω αγγλικά, μη βάλετε ακουστικά. Πολλές θεμι... Οι ερωτήσεις είναι θεμητές. Είπατε ότι ως Ευρωομάδα θα δουλέψουμε πολύ τους επόμενους μήνες και ιδιαίτερα τον Νοέμβρη για τις συστάσεις για κάθε χώρα, σχέδια προϋπολογισμών και με τις απόψεις της Κομισιόν ε, πάνω σε αυτά και θα δώσουμε συμπεράσματα από τις συζητήσεις μας τον Νοέμβριο. Για την Τραπεζική Ένωση. Τα περισσότερα δομικά στοιχεία της Τραπεζικής Ένωσης συζητούνται στο ΕΚΟΦΗΝ βέβαια μεταξύ της Προεδρίας και ε, του Κοινοβουλίου και του ΕΚΟΦΗΝ. Η... Όμως τα συμφέροντα της Ευρωομάδας είναι πολύ κέρια εδώ, οπότε θα υπάρχει πολύ στενή συνεργασία μεταξύ ΕΚΟΦΗΝ και Ευρωομάδας. Θα ζητήσουμε από την ΕΚΤ και τον Πρόεδρό της να μας ενημερώσει για το πώς η ΕΚΤ θέλει να οργανώσει τη διαδικασία της αξιολόγησης των ισολογισμών και νομίζω ότι η καθαρότητα, η σαφήνεια για όλους τους ενδιαφερομένους και τους υπουργούς και του κόσμου είναι σημαντική. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, να πιστεύουν όλοι ότι η διαδικασία είναι καλή, σωστή, ότι θα γίνεται με τρόπο ανεξάρτητο και με τρόπο πολύ ποιοτικό. Δεν ξέρω ποια χρονική στιγμή ο πρόεδρος της ΕΚΤ θα μας ενημερώσει για την οργάνωση όλου αυτού του εγχειρήματος, υποθέτω σύντομα. Τώρα, από αυτή τη διαδικασία το συμπέρασμα μπορεί να είναι ότι μπορεί να χρειάζονται κάποιες τράπεζες σε περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση. Η συνήθι σειρά, η ακολουθία είναι πρώτα η τράπεζα να ψάξει από τις κεφαλαιαγορές να βρει λεφτά, κονδύλια ή από την αναδιάρθρωση της επιχείρησης, οπότε πρώτα είναι ευθύνη της τράπεζας να τα φροντίσει αυτά, πριν μιλήσουμε για χρήση δημοσίων κονδυλίων και μέσων προστασίας. Θα πρέπει να ισχύσουν και οι κανόνες κρατικής ενίσχυσης ε, και θα πρέπει ίσως να γίνει και μια, ένα μπεϊλίν, εσωτερική διάσωση. Μετά θα υπάρξουν, ε, σε κάποιες χώρες υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για την εξυγίανση, μπορεί να υπάρξουν προστατευτικοί μηχανισμοί εθνικοί αν χρειαστεί, αλλά όλα αυτά είναι στην μεταβατική φάση. Η χρήση άμεσα ανακεφαλαιοποίηση αυτή τη μεταβατική φάση, αυτή τη φάση της αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων θα είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει για παράδειγμα μια προϋπόθεση για την ε, άμεση, ε, χρήση κονδυλίων άμεσης ανακεφαλαιοποίησης από τον ESM θα ε, γιατί έχει, ότι θα έχει αρχίσει το εποπτικό έργο της ΕΚΤ και δεν θα έχει αρχίσει μέχρι κάποιους μήνες, οπότε υπάρχει θέμα χρονικής στιγμής αν και όποτε γίνει άμεση ανακεφαλαιοποίηση σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, ε, υπάρχουν και συγκεκριμένοι όροι, μια σειρά όρων. Ένας άλλος όρος είναι ότι ε, το, θα πρέπει να έχει εξαντληθεί το, και θα εφαρμόζεται το εσωτερικό κούρεμα, το bail όπως λέμε, από το, με βάση την οδηγία για την εξυγένση και ανάκαμψη των τραπεζών. Ε, υπάρχουν δηλαδή, προβλέπεται, αλλά υπάρχει μια αυστηρή αιρεσιμότητα, δηλαδή προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν. Ευχαριστώ. Νομίζω αυτό μα δίνει αφορμή για να έχουμε στη συνέχεια και επιπλέον ε, ερωτήσει για το ίδιο θέμα. Η Ελίζα Φεραίρα για του σοσιαλιστέ. Θα μιλήσω πορτογαλικά, με συγχωρείτε, βάλτε τα ακουστικά σα. Ευχαριστώ πολύ που και πάλι είστε εδώ μαζί μας. Περνάει και ώρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε και πάλι εδώ μαζί μας. Η ερώτησή μου αφορά τη νέα φάση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Νέες απαιτήσει για τις χώρες, αλλά πράγμα που επιφέρει και περισσότερες ευθύνε, διότι θα πρέπει να υλοποιήσουν τις συστάσεις. Στην πραγματικότητα ως τώρα βλέπουμε οι συστάσεις που έχουν ε, διατυπωθεί, να μην έχουν επιτύχει τους ε, επιδιωκόμενους στόχους. Διαρκώς υπάρχει ε, πρόβλημα με τις εκτιμήσεις και για την ανάπτυξη και για το χρέος και για την απασχόληση και αυτό βεβαίως είναι ένας παράγων ο οποίος ε, ουσιαστικά ε, απογοητεύει τις χώρες που σε πολλές περιπτώσεις έχουν ακολουθήσει κατά γράμμα τις συστάσεις Σήμερα λοιπόν δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τις προπτικές ανάπτυξης των διάφορων οικονομιών, κάτι που θα μπορούσε να γίνει εάν ήταν εκτιμήσει διαφορετικές αλλά τελικά ζουν την ύφεση λόγω των συστάσεων. Ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξή. Με τις νέε αρμοδιότητες που θα σα ανατεθούν θα υπάρχει περισσότερο προσεκτική ε, αξιολόγηση των ε, συστάσεων οι οποίε μετά επιβάλλονται στις διάφορες χώρες και προκειμένου να επιδείκονται πραγματικά αποτελέσματα, όχι θεωρητικά. Αυτά όλα προκαλούνται από τις συστάσεις που εικονείται. Θα υπάρχει μια εντελεχής ανάλυση της, της εσωτερικής ζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί την ώρα απασχολούμαστε με την προσφορά περισσότερο και όχι με την ζήτηση. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως αυτές ε, της ζώνης ευρώ, του ενιαίου οικονομικού χώρου, ε, έχουν, ε, υλοποιούν αυτή τη στιγμή πολιτικές ύφεση. Κάτι που δεν επιτρέπει την τόνωση τη ζήτηση. Σε ένα-δύο χρόνια ε, όλη η παραγωγική δομή τη εσωτερική αγορά θα έχει καταρρεύσει και θα έχουν όλα εξαχθεί προ την ε, διεθνή αγορά. Άρα το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να είμαστε λιγότερο συναισθηματικοί και λιγότερο ε, δραματικοί στην προσέγγιση μας και να είμαστε περισσότερο πραγματιστές στην εκπόνηση των συστάσεων. Αυτή η πρώτη ερώτηση και η δεύτερη για να ρωτήσω σε σχέση με τα χρέη των κρατών. Το πρόβλημα δεν έχει επιληθεί. Ας δούμε την Ελλάδα. Ελλάδα. Το χρέο έχει αυξηθεί διότι υπάρχει εσωτερική ύφεση και το χρέο πολλαπλασιάζεται. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να τροποποιηθεί, να μεταβληθεί η στάση σα. Υπάρχει μια μέρημνα και για την κοινωνική διάσταση. Κάτι ελάχιστο για να λάβουμε υπόψη και τι δαπάνε και την κάλυψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που σχετίζονται ακριβώ ε, με του πολίτε και οι οποίοι πρέπει να υποστούν τι πολιτικέ λιτότητε οι οποίε έχουν οδηγήσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ, κύριε Φεραίρα, για την ερώτησή σας. Η πρώτη σας ερώτηση αφορά την ποιότητα των συστάσεων. Οι συστάσεις συζητήθηκαν στο Eurogroup πριν το καλοκαίρι και δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι οι προηγούμενες συστάσεις δεν ήταν καλής ποιότητας. Και αυτό γιατί δεν έχουμε διαφύγει πλήρως από την κρίση. Όχι, κινούμαστε αργά-αργά εκτός του πλαισίου της ύφεση, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς και να πούμε ότι η οικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν βαθύτερη και δυσκολότερη να αντιμετωπιστεί από ό,τι υπολογίζαμε αρχικά. Όμως σιγά σιγά κινούμαστε μακριά από την ύφεση σε πολλές χώρες. Δεν μπορείτε λοιπόν νομίζω να πείτε ότι ήταν εσφαλμένες οι κινήσεις μας. Πολλέ από τι μεταρρυθμίσει ήταν απαραίτητε σε πολλέ από τις χώρες. Μεταρρυθμίσεις ανά χώρα διαφορετικές βέβαια, αλλά οι περισσότερες σκοπό έχουν να εξυγχρονίσουν την οικονομία, να κάνουν ανταγωνιστικότερε τι οικονομίε τη κάθε χώρα και όλε αυτέ οι μεταρρυθμίσει πρέπει να προχωρήσουν θα μπορούσε κανεί να προβάλλει το επιχείρημα ότι δεν έχει επιτελεστεί αρκετή πρόοδο. Αλλά γι' αυτό δεν φταίει η ποιότητα των συστάσεων, αλλά η ποιότητα τη υλοποίηση των συστάσεων αυτή καθ' αυτή. Το τι πρόοδο έχουν επιτελέσει οι ίδιε οι χώρε. Αυτό μας έχει απασχολήσει και από τεχνικής άποψης βεβαίως έχει επιτελεστεί πρόοδος. Τα ελλείμματα στον προπολογισμό έχουν ε, μειωθεί σε πολλές χώρες, έχουν περιοριστεί. Και όπως ορθώς είπατε, το κοινωνικό τίμημα ήταν σαφώς βαρύ, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι το τελευταίο εξάμεινο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιτρέψει, έχει δώσει περισσότερο χρόνο στι περισσότερε χώρε, ιδίω την απάντηση στι διάφορε συστάσει, την απάντηση πρέπει να ξέρουν στι διάφορε συστάσει και λόγω τη ύφεση. Έχουν λοιπόν περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στου δημοσιονομικούς στόχου. Αυτό ήταν μια αλλαγή στη διαδικασία των συστάσεων, στη διαδικασία των στόχων που τίθενται για το σκέλο του δημοσιονομικού ελλείμματο. Το τελευταίο ερώτημα σα αφορούσε το χρέο. Το χρέο είναι κάτι που πολλαπλασιάζεται βεβαίω διαρκώ σε περίοδου κρίση και είναι πολύ δύσκολο κανεί να το ξεφορτωθεί και να το περιορίσει. Αυτό ισχύει για πολλέ από τι χώρε μα. Ε, το χρέο είναι υψηλό και το αναμέναμε αυτό ακόμα και στι χώρε που βρίσκονται στο πλαίσιο τη Τρόικα. Πολύ αργή είναι η διέξοδο από την κρίση και την ύφεση για τι χώρε αυτέ. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην ποιότητα των συστάσεων. Περισσότερο στην ποιότητα τη υλοποίηση των ταπέδιδα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση, κυρία Γκουλάρ, για του φιλελεύθερου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Εκτίμησα ιδιαίτερα αυτό που είπατε και θα συμφωνήσω με αυτό που είπε και η Κορίν Κόλ. Δεν σημαίνει ότι επειδή συμμετείχαμε στην νομοθετική διαδικασία. Μ' ακούτε? δεν σημαίνει ότι η υλοποίηση πρέπει να γίνει όπως έχει ακριβώς προβληθεί. Και στο παρελθόν είχαμε πρόβλημα υλοποίησης ε, με τους κανόνες που είχαμε αποφασίσει από κοινού. Το Eurogroup νομίζω έχει έναν καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει εδώ. Διότι σε κάποιες χώρες, εκ των οποίων και η Γαλλία δυστυχώς, υπάρχει τάση να λέμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπαγορεύει πράγματα στις χώρες. Όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπέρμετρε αρμοδιότητε. Όμω αυτέ οι αρμοδιότητε έχουν χωρίσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι ο ρόλο τη. Άλλωστε και εμεί θεωρούμε ότι το ρόλο αυτό τον εκτελεί με ίσως μεγαλύτερη κριτική ικανότητα από ό,τι στο παρελθόν και μεγαλύτερη ευθύνη. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι τεχνικό, είναι πολιτικό. Πρέπει να δείξουμε στου πολίτες της Ευρώπη ότι αυτέ οι κοινέ διαδικασίε έχουν κάποια σημασία και νόημα. Και μια άλλη παρατήρηση είναι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Όλες οι προτεραιότητες που έχετε θέσει είναι ευστοχές και αποδοτικές, όμως με τρομάζει που η ενέργεια των νέων φτάνει, έρχεται τελευταία. Γιατί, διότι αν χάσουμε την νεολαία μας, ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε κατά τα άλλα, θα θεωρηθεί ως αθέμητο και θα το πληρώσουμε στις επόμενε ευρωεκλογέ. Άρα, ίσως και να είναι θέμα της παρουσίαση, αλλά ίσως όχι μόνο, να είναι και θέμα διάρθρωσης και μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Τι μπορείτε να κάνετε στην πράξη, τι έχετε την πρόθεση να κάνετε για να καταπολεμήσετε τον κατακαιρματισμό της αγοράς ως προ τα επιτόκια. Διότι όχι μόνο υπάρχουν ε, αποκλήσει και διαφορέ, όπω είπατε, αυτό στην πραγματικότητα μεταφράζεται με ε, δυσκολίες ανταγωνιστικότητας, διακοπές ανταγωνιστικότητας εντός στην εσωτερική αγορά. Προφανώς αυτό χρειάζεται επεξεργασία, αλλά τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει στην πράξη από λειτουργικής πλευράς για να αντιμετωπιστεί αυτό. Ευχαριστώ. Μάλλον έχετε δίκιο. Το Eurogroup έχει σημαντικό ρόλο εδώ να διαδροματίσει και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο επίση και στον τρόπο που οι συστάσεις διατυπώνονται. Και μετά στο πώ υλοποιούνται. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Αυτό ακριβώ είναι ο ρόλο που θέλουμε και να, έχουμε, και να διαδραματίζουμε. Στη συζήτηση τώρα που προέκυψε μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γαλλία, να πω ότι για οποιαδήποτε χώρα ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να αναλύσει ποια είναι τα διαφορετικά προβλήματα τη οικονομία και τι εμποδίζει την ανάκαμψή τη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα μπορεί να συστήσει μέτρα για την αγορά εργασία, λόγω χάρη, εφόσον εκεί εντοπίσει προβλήματα, εφόσον εκεί υπάρχουν ανεπάρκειε ο τρόπος που ε, στην πράξη κάθε χώρα θα αποφασίσει να λύσει το πρόβλημα, αυτό μπορεί να το αποφασίσει η ίδια η χώρα κατά μεγάλο μέρος. Έτσι και θα πρέπει να συνεχίσουμε. Εάν έβλεπε, αν έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάντε αυτό ή εκείνο, ας πούμε αλλάξτε το συνταξιοδοτικό σας σύστημα, νομίζω ότι η χώρα σε εθνικό επίπεδο και αυτό είναι και θέμα δημοκρατικής νομιμότητας, θα έπρεπε να αποφασίσει με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει εντοπιστεί. Έπειτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurogroup θα μπορούσαν να αποτιμούν κατά πόσον τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν επαρκή για να αντιμετωπιστεί το διαφορετικό πρόβλημα. Αυτό είναι ο σωστό τρόπο. Έτσι θα έπρεπε να γίνεται η όλη διαδικασία. Είναι σαφέ λοιπόν η Γαλλία, και αυτό ισχύει για οποιαδήποτε άλλη χώρα, η Γαλλία οφείλει κάτι τέτοιο να κάνει. Το πώ ακριβώ όμω θα το αντιμετωπίσει το διαφορετικό πρόβλημα, αυτό είναι δικό τη θέμα, κατά πρώτο λόγο. Είναι δική τη ευθύνη και θα αποτιμηθεί εκ των υστέρων. Για την νεολαία και την ανεργία. Ως πολιτικός άντρα κι εγώ ήξερα από ανέκαθεν, ήξερα μάλλον ανέκαθεν ότι αν θέλετε ένα θέμα να είναι πολύ κάτι που θα μείνει στο νου των ακροατών σα, είναι κάτι που να αναφέρεται στο τέλος. Γι' αυτό αναφέραμε την, την ανεργία των νέων τελευταία, γιατί είναι το πλέον σημαντικό. Οι διαρθρωτικέ αλλαγέ στην οικονομία μα, με τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τι διαρθρωτικέ δυσκολίε, όλα στο τέλο οδηγούν έναν βασικό στόχο, την οικονομική ανάκαμψη όσο το γρηγορότερα, ώστε να μπορέσουν να έχουν νέε ευκαιρίε για νέε θέσει εργασία. Υπάρχει ένα άμεσο τρόπο να αντιμετωπιστεί αυτό, γι' αυτό και διατίθενται κονδύλια, υπάρχουν προγράμματα που εκπονούνται για του νέου, το Ταμείο για την Ανεργία των Νέων, γι' αυτό προέκυψε αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων. Και είναι ένα περισσότερο μακροοικονομικό τρόπο για να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να δούμε τα δομικά ε, προβλήματα τη οικονομία μα και πώ θα μπορέσει να επανέλθει αύξηση και ανάπτυξη για του νέου. Και για τον κατακαιρματισμό των αγορών. Το ίδιο θα πω και εδώ. Υπάρχει ένα τρόπο πιο βραδύ να αντιμετωπιστεί το θέμα ή έστω πιο, έστω πιο μεσοπρόθεσμο, η εστω πιο Ένωση. Αλλά δεν λειτουργεί ακόμη διατραπεζικά το σύστημα των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των χωρών. Υπάρχει κατακαιρματισμό. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη, οι μένε στι τράπεζε των ΔΕ, και να ε, αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία των τραπεζών. Η Τραπεζική Ένωση αυτό είναι επιδιώκει και γι' αυτό βιαζόμαστε τόσο και θέλουμε να καλύψουμε όλα τα στοιχεία τη. Ο πιο σύντομο τρόπο να γίνει κάτι τέτοιο είναι απλώ να έχουμε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ώστε να διατεθούν κονδύλια για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Σε αρκετέ χώρε υπάρχουν εθνικέ πρωτοβουλίε σχετικά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διδραματίζει ένα ρόλο εδώ, αλλά αν όλα πάνε καλά, σύντομα θα έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα με τη συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Έχουμε πέντε λεπτά, δεν τα πάμε πολύ καλά. Είναι συλλογική η ευθύνη μα εδώ για του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, ο κύριο Βαντάλμεν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα το πρωί κύριε Ντάιζελμπλουμ. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο πολύ δύσκολο έργο σα. Υπάρχουν ε, κάποιες συστάσεις αναχώρα στις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ. Πρώτα απ' όλα, ό,τι αφορά την Ελλάδα, είπατε ότι στο μέλλον θα δοθεί ένα νέο δάνειο στην Ελλάδα. Τι είδους δάνειο θα είναι αυτό όμως θα είναι ένα δάνειο που θα χρησιμεύσει για την εξυπηρέτηση προηγουμένων δανείων ή θα είναι ένα δάνειο το οποίο στόχο θα έχει ε, την μείωση του πραγματικού χρέους ε, στην χώρα, εντός της χώρας. Και το δεύτερο μου ερώτημα είναι το εξής. Ακούμε κάποιες παλιές καινούριε ειδήσει. Ε, τελικά κάποιες φορές δεν πρόκειται καν για είδηση. Άλλες φορές δεν ακούμε κάτι καινούριο. Το θέμα να δούμε τι μέλη γενέστε. Ο οικονομολόγος Χράβελαντ μιλάει για την ε, αποσταθεροποίηση στη Γερμανία και λέει ότι καλό θα ήταν να παραγραφεί ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέους. Αν μιλάμε για νέο υποτιμένο νόμισμο. Ίσως αυτό θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερες ελπίδες και περισσότερες δυνατότητες. Όλα αυτά, αυτή τη δήλωση τέλο πάντων του οικονομικού αυτού, πώς την κρίνεται. Επίσης, Λάβαμε κάποια έγγραφα για τη σημερινή συνεδρίαση. Μεταξύ αυτών, το Ινστιτούτο Μπρούκελ μιλάει για ένα negative output gap. Ε, Ιταλία, Ολλανδία έχουν δυσκολίες τι θα πει αυτό όμως ακριβώς. Αν αυτό το παραγωγικό κενό, το παραγωγικό χάσμα, το αρνητικό συνεχίσει να διευρύνεται, τι επίπτωση θα έχει αυτό. Τι δομικές πτυχές ενδεχομένως θα περιλαμβάνει. Μήπως έχει αντίκτυπο και στην ανεργία. Από την ιδιότητά σας λοιπόν ως επικεφαλής του Eurogroup Μήπως θα μπορούσατε ενδεχομένως να προσεγγίσετε τον Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών. Μήπως θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τις επενδύσεις, να κάνουμε κάτι για την αντιμετώπιση της λιτότητας. Απάντησα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας κύριε Φαντάλεν που βέβαια κατά κύριο λόγο μιλούσε για την Ελλάδα και είπατε νέο δάνειο για την Ελλάδα. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι μετά το τέλος αυτού του προγράμματος, του τρέχοντος, υπάρχουν λόγοι που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν θα έχει εντελώς βγει από την προβληματική θέση στην οποία βρίσκεται τώρα η Ελλάδα και ότι θα χρειαστεί μάλλον περαιτέρω βοήθεια. Ίσως θα είναι απαραίτητη περαιτέρω βοήθεια. Πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα, να είμαστε σαφείς. Από τότε που εγώ ε, έγινα μέλος του Eurogroup πάντα λέγαμε ξεκάθαρα ότι ακόμη και μετά το τέλος ε, του προγράμματος αυτού μέχρι το 2014 εάν χρειαστεί ε, περαιτέρω βοήθεια ή είμαστε έτοιμοι Europe τα λοιπά Έτσι κάπως το διατύπωσα. Δεν ε, υπάρχει είδηση εδώ, ε, καμία νέα είδηση και νομίζω ότι αυτό ήταν και το δεύτερο. Πόσο καιρό ακόμα θα ακούμε αυτές τις ειδήσει που δεν είναι ειδήσει πια. Είπαμε ότι θα βοηθήσουμε την Ελλάδα μέχρι να σταθεί στα πόδια της και να ε, έχει πλέον πάλι πρόσβαση στις αγορές. Αλλά είπαμε ότι πρέπει η Ελλάδα να εξακολουθήσει να εκπληρώνει όλους τους όρους του μνημονίου. Επίσης μου αναφέρατε αυτή την έκθεση που λέει για το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Εγώ πρέπει να σας πω ξεκάθαρα ότι υπάρχει ομοφωνία εντός του Eurogroup ως προς το ότι η Ευρωζώνη, η ακαιρεότητα της Ευρωζώνης ε, θα παραμείνει ανέπαφη. Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι να βοηθήσουμε τις χώρες που χρειάζονται βοήθεια και στήριξη εκεί που τη χρειάζονται και δεν θα συζητήσουμε τίποτα. Ε, δεν είναι υποσυζήτηση καν το θέμα της ακαιρεότητας της Ευρωζώνης. Ό,τι αφορά την υποτίμηση, η υποτίμηση δεν αποτελεί μέθοδο, ανεξαρτήτως των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων που θεωρείται ότι έχει, η υποτίμηση όμως δεν είναι ένα μέτρο για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων τη ανταγωνιστικότητας και άλλων διαρθρωτικών προβλημάτων ε, των οικονομιών. Είναι ένας τρόπος να παρακάμψουμε το πρόβλημα, αλλά όχι να το αντιμετωπίσουμε. Τέλος, νομίζω το ερώτημά σας αφορούσε το τελευταίο, δηλαδή την εσωτερική Ολλανδική πολιτική, ε, αν θα πρέπει να γίνουν περικοπές ή όχι. Εγώ ως Ολλανδός υπουργό, δεν θέλω βέβαια να ε, αποφύγω να απαντήσω, ούτε να επεκφύγω. Θα υπάρξουν ε, περικοπές, θα γίνουν μακρές συζητήσεις για μεταρρυθμώσεις βέβαια, αλλά θα υπάρξουν και περικοπές. Απλά και μόνο για να τηρήσουμε τους κανόνες, να εφαρμόσουμε και εμείς τους κανόνες που έχουμε θέσει για όλες τις χώρες. Δεν ισχύουν για τι άλλε χώρε μόνο, ισχύουν για την Ολλανδία αυτοί οι κανόνες. Και τώρα για του πρασίνους ο Σβέν Γκίγκολτ. Κατά πρώτον, ευχαριστούμε που ήρθατε και πάλι. Και ελπίζουμε ότι περάσετε ωραίε διακοπέ. Θα το χρειαστείτε. Εάν σκεφτούμε πώς θα πρέπει να υλοποιήσετε τα θέματα της Τραπεζικής Ένωσης. Κάτι που προφανώς είναι το σημαντικότερο βήμα που πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Ακόμα και αν υπάρχουν δυσκολίε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι διαπραγματεύσει σχετικά, ε, είμαστε στη διαδικασία τη ε, περάτωσης της νομοθετικής διάστασης. Το βασικότερο εδώ θα είναι η υλοποίηση όμω. Ακούω κάποια σχόλια και κάποια από αυτά που ακούω τα βρίσκω ανησυχητικά. Η ρυθμιστική διάσταση λέει διάκριση των δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο φρόντισαν να υπάρχει ισχυρή, ισχυρός πρόεδρος για το Συμβούλιο Εποπτών. Ε, στο ενδιάμεσο όμως. Ποιος θα ελέγχει, ποιος έχει τον έλεγχο, πώς θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι το Συμβούλιο των Εποπτών θα αρχίσει να εργάζεται γέρος και αυτό στα τα δημοκρατικά δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την δημοσιονομική πολιτική να μην πληγούν de facto λόγω της προπαρασκευαστικής περίοδου. Και τα βασικά στοιχεία του πλωστασίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Εποπτικού του Συμβουλίου να υπάρχουν και να λειτουργούν εγκαίρως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι το πρώτο που έχω να πω. Και κατά δεύτερον, όταν προβλέψατε την Τραπεζική Ένωση, θεωρήσατε ότι χρειάζονται εκθέσεις ε, αξιολόγησης, ποιοτικέ. Αν αυτό συμβεί, θα πληγεί, δεν συμβεί, θα πληγεί το κύρος της, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όμως το βασικό ερώτημα είναι το εξή και αυτό το είπαν και οι πυρογνώμονες. Αυτοί οι πυρογνώμονες, από πού θα προέρχονται, από τις αρμόδιες αρχές των εθνικών κρατών, από τις τράπεζές τους, θα ετοιμάζουν ε, την εξέταση, την έκθεση για τα περιουσιακά στοιχεία ε, τη τράπεζας. Αυτή είναι εξάρτητη εμπειρογνώμων στην τομέα συμπεριλαμβανομένων και των υπευθύνων για τη σύνταξη των ε, εκθέσεων περιουσιακών στοιχείων ε, των τραπεζών των κατώμελών μέσα από το νέο τραπεζικό σύστημα. Ευχαριστούμε κύριε Γκίγκολτ για τις ερωτήσεις σας. Η υλοποίηση είναι όντως ζωτική σημασίας και από την άποψη των συγκεκριμένων συστάσεων για τις χώρες αλλά και από την άποψη της Τραπεζικής Ένωσης. Ως προς τις ανησυχίες σας, τέλος πάντων τις αμφιβολίες σας για το Εποπτικό Συμβουλίο και το κατά πόσον αυτό θα μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι της δουλειάς μας και κατά πόσον θα είναι και ανεξάρτητο από την πλευρά των υπερογνωμόνων, εδώ συμφωνήσαμε Ε, με την πρόταση για τις ε, για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, το Εποπτικό Συμβούλιο να ξεκινήσει ένα χρόνο μετά την δημοσίευση της πρώτης έκθεσης. Η δημοσίευση αυτής, αυτής της πρώτης έκθεσης επίκειται. Πολύ σύντομα θα την έχουμε. Οπότε θα υπάρχει ένας χρόνος για όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες. Αλλά και προηγουμένως πριν την επίσημη αρχή του ε, λειτουργίας του Ενίου αποπτικού μηχανισμού θα πρέπει να υπάρξει και ενημέρωση του ΕΚΟΦΗΝ. Ε, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ενημερώσει το ΕΚΟΦΗΝ για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις προετοιμασίες μας. Ένα από τα βασικά ζητήματα εδώ είναι το Εποπτικό Συμβούλιο να είναι πανέτοιμο για να αναλάβει τις αρμοδιότητές του. Προφανώς αυτό πρέπει να γίνει ε, και να γίνει στα πλαίσια της ανεξαρτησίας που λέγατε. Ε, για την αρχή λειτουργίας, την επίσημη αρχή λειτουργίας του εποπτικού μηχανισμού το φθινόπωρο το 2014. Έχουμε όμω ένα χρόνο. Και όσο αφορά του ανεξάρτητου εμπρευνόμονε και τι ιδιωτικέ εταιρείε για τη διαδικασία αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, ε, δεν μπορώ εδώ να τοποθετηθώ. Έχω ξαναδηλώσει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει εντελεχής και ανεξάρτητη μελέτη και ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού ω μέρο των εκτίσεων αυτών. Οι ιδιωτικέ εταιρείε πρέπει εδώ να αναλάβουν κάποιο ρόλο σίγουρα και αυτό το θεωρώ απαραίτητο. Για τι λεπτομέρειε όμω τη πρακτική διοργάνωση αυτού του θέματο, αυτά δεν έχουν ακόμη εξεταστεί πλήρω. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μα ενημερώσει και από την πλευρά του ΕΚΟΦΗΝ και από την πλευρά του Eurogroup και συμφωνώ απολύτω μαζί σα. Πρέπει να υπάρχουν τα ύψιστα δυνατά πρότυπα. Okay, ε, Εντάξει. Ο κύριο Φουντή για την ΚΟΕ. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με προσοχή αυτά που μας είπατε εισαγωγικά Άκουσα με προσοχή τις αναφορές σας στο ελληνικό πρόγραμμα και επίσης και τις απαντήσεις σε προηγούμενες ερωτήσεις των συναδέλφων. Θέλω να σας πω ότι για τις εκτιμήσεις σας για το ελληνικό πρόγραμμα επισκεφτήκατε και την Ελλάδα και τα λοιπά, δεν συμφωνώ ε, και δεν συμφωνούν μαζί σας κατά τη γνώμη μου και τα στοιχεία τόσο για την πορεία του χρέους όσο και για την πραγματική οικονομία, ανεργία και ούτω καθεξής. Ισχυριστήκατε σε σχετική ερώτηση ότι δεν φταίει η συνταγή, δεν φταίει το σχέδιο, αλλά φταίει η εφαρμογή. Ας πάμε τώρα λίγο στην εφαρμογή για να σας πω τι θέλω να σας ρωτήσω για να μου το διευκρινίσετε. Επανειλημμένα και σήμερα και σε γράμμα που στείλατε στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο μιλήσατε ότι το πιο πιθανό είναι η Ελλάδα δεν θα βγει στις αγορές το 2014 και θα χρειαστεί ένα νέο πακέτο βοήθειας με πρόσθετους επαρκείς όρους. Επειδή η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων πολιτών έχει κάποια όρια, το ίδιο και οι μεταρρυθμίσεις, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ασκείτε κριτική και σήμερα νομίζω και στην τοποθέτησή σας υπονοήσατε ότι δεν προχωράνε οι μεταρρυθμίσεις, υπάρχει πρόβλημα μεταρρυθμίσεων ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα. Ασκείται κριτική ότι δεν προχωράει αυτό το πρόγραμμα επαρκώς. Η ερώτηση λοιπόν κύριε Πρόεδρε έχει να κάνει με το εξή. Μέσα στο πλαίσιο της παρακολούθησης των μεταρρυθμίσεων που γενικώ μας είπατε και ειδικά για την Ελλάδα. Πρώτη ερώτηση. Υπάρχουν σκέψεις στο Eurogroup ή στο ESM για στενότερο έλεγχο των μεταρρυθμίσεων και ειδικά των ιδιωτικοποίησεων στην Ελλάδα έχουμε διαβάσει διάφορες δηλώσεις. Και το δεύτερο συμπληρωματικό, σε αυτούς τους πρόσθετους όρους με τους οποίους θα δοθεί κατά πάσα πιθανότητα νέο πακέτο βοήθειας υπάρχει και αυτή η πλευρά, δηλαδή ότι εσείς οι δανειστές συγγνώμη, θα παρακολουθούν πιο στενά τις μεταρρυθμίσεις και ιδιαίτερα τις ιδιωτικοποίησεις στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Χούντι για τις ερωτήσεις σας. Οι παρατηρήσεις μου σχετικά με την εφαρμογή αφορούσαν ειδικά τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εις ό,τι αφορά προϋπολογισμό και ελλείμματα, αυτό αφορά πάρα πολλές χώρες. Οι στόχοι έχουν επιτευχθεί ή προσαρμοστεί ε, θετικά λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ύφεση και τις κοινωνικές επιπτώσεις κάποιων δημοσιονομικών στόχων. Από την πλευρά του προϋπολογισμού λοιπόν δεν ε, επικρίνω την εφαρμογή. Από την άποψη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων βλέπω και το βλέπω και από το εθνικό επίπεδο ότι είναι πολύ δύσκολο να σπρώξουν κάποιες μεταρρυθμίσεις απαραίτητες. Καμιά φορά είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει απαραίτητη πολιτική υποστήριξη κλπ. Ναι, εις ό,τι αφορά την εφαρμογή με απασχολούν λοιπόν και ανησυχώ σχετικά με την ταχύτητα εφαρμογής και τα παραδοτέα στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αλλά αυτό είναι πιο γενική παρατήρηση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Τώρα, για πρόσθετες προϋποθέσεις για την Ελλάδα, πρόσθετους όρους. Είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, για να μιλήσουμε για τον χαρακτήρα ενός νέου προγράμματος, το μέγεθος ενός πιθανού νέου προγράμματος ή τους όρους ενός νέου προγράμματος. Δεν μπορώ να επισέλθω εδώ. Το μόνο που ξεκαθάρισα πολλές φορές είναι ότι είναι πολύ πιθανό στο τέλος αυτού του προγράμματος να χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση η Ελλάδα και τα προβλήματα της Ελλάδας δεν θα έχουν επιληθεί και ότι δεν θα υπάρχει στο τέλος του 2014 επίτευξη πλήρους πρόσβασης στις αγορές. Και το, η Ευρωμάδα είναι έτοιμη να παράσχει περαιτέρω βοήθεια και στήριξη στην Ελλάδα όποτε χρειαστεί κλπ. Αυτή είναι η στάση μου, αυτή είναι η θέση μας. Αυτά είναι όσα συμφωνήσαμε στη δήλωση του Δεκεμβρίου της Ευρωομάδας. Αλλά το ποια θα είναι η υποστήριξη, η βοήθεια που θα δοθεί στην Ελλάδα μετά το 2014, δεν μπορώ να σας το πω. Είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς για τέτοιου είδους εικασίες. Τώρα για τις μεταρρυθμίσεις ε, και αν θα πρέπει να εποπτεύονται ή να παρακολουθούνται ακόμα πιο πολύ. Γενικά οι ε, και το πλάνο για τι μεταρρυθμίσει για την Ελλάδα είναι σαφές. Υπάρχουν μεγάλα θέματα, μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Άσχετα από το αν είναι σε κρίση ή όχι μια χώρα, ένα αποτελεσματικό σύστημα φορολογικό, αποτελεσματικό, αποδοτικό, αυτό είναι κέρια σημασία για κάθε χώρα που θέλει να διατηρήσει το κοινωνικό τη σύστημα και την εθνική τη οικονομία υγιή. Οπότε εκεί ε, πολλή δουλειά μπορεί να γίνει και πολλοί βοηθούν στην Ελλάδα για να εφαρμοστούν αυτές οι συστάσεις. Ευχαριστώ. Πρέπει να επιταχύνουμε όμως γιατί θα δυσκολευτούμε με τις επόμενες ερωτήσεις. EFD, ε, Bastian Belder. Σας ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε του Γιώργου, κύριε Ντάιζελ Μπλουμ. Η Ευρωζώνη έχει να αντιμετωπίσει μια τεράστια πρόκληση, διότι Έχουμε τεράστιο ε, χρέος, ε, ε, θέμα ανταγωνισμού μεταξύ χαρών, μάλλον μείωση της ανταγωνιστικότητα σε πολλές χώρες. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει πρόβλημα και με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες στην Ένωση και δεν θα πρέπει να την θέσουμε σε κίνδυνο αυτή την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει κάτι να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε ε, στον ε, κόσμο. Το να μιλάμε για λογαριασμούς, να μιλάμε για ε, πληθωρισμό. Το θέμα δεν είναι αυτό ακριβώς, είναι να ξέρει ο κόσμος τι μπορεί να περιμένει για το μέλλον και τι είδος δίκτυα ασφαλείας μπορεί να υπάρξει για πιο αδύναμες τράπεζες ή να δούμε τι γίνεται με τις τεράστιες ανισορροπίες, πώς μπορούμε να έχουμε μια μακροχρόνια αναχρηματοδότηση σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση. Θα πρέπει να δοθεί κάποια κεφαλαιανική ενίσχυση στις ε, τράπεζες σε εθνικό επίπεδο και αυτό πάνω με φαίνει στην πρώτη μου ερώτηση. Νομίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, επαρκή περιθώρια για να μπορούν να προβούν σε ανακεφαλοποίηση των τραπεζών τους στη χώρα από μόνες τους και αν όχι οι χώρες που έχουν ήδη ξεκινήσει την αναδιάρθρωση ε, του τραπεζικού τομέα, Ολλανδία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε ξεκινήσει εκεί τις προσπάθειες για την εξήγηση των ισολογισμών. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχει στον αντίποδα πρόβλημα σε πολλές άλλες ε, χώρες. Τι γίνεται με αυτό. Τρίτον, Τι θα γίνει με την Τραπεζική Ένωση αν έχουμε τεράστιες ε, απώλειες. Πώς θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, σε ερωτήσεις σας κύριε Μπέλτρικ, και ο Σντάιζελμπλουμ. Η Τραπεζική Ένωση, ξέρετε, δεν είναι ε, η Πανάκια είναι για όλα. Θα είναι ένα σύστημα που θα μας βοηθήσει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ τραπεζών και στις τράπεζες. Και δεν θα δοθούν λευκές επιταγές σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε αυτό το νέο εγχειρίδιο κανόνων, το Single Rulebook και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και σχετική οδηγία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Οι τράπεζες πλέον όλες θα πρέπει να ε, έχουν ποιοτικού ισολογισμούς. Δεν είναι κάτι που μέσα σε μια χρονιά θα το επιτύχουν, έχουν ε, κάποια χρονική προθεσμία, αλλά οι χρηματοπιστωτικέ αγορές πιέζουν και οι ρυθμιστές και οι ΕΚΤ θα πιέσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Έπειτα, Έχουμε τον νέο εποπτικό μηχανισμό. Η ΕΚΤΑ σε συνεργασία με τους εθνικούς επόπτες θα καταβάλει προσπάθειες ώστε οι τράπεζες να γίνουν υγιείς, να είναι ευρωστές να αρχίσει να κινείται πάλι ο τραπεζικός τομέας. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της ΕΚΤ λοιπόν. Εσείς όμως λέτε τι θα γίνει αν ε, προκύψουν νέα προβλήματα στις τράπεζες ε, και ε, κάνετε κάποιες υποθέσεις που δεν με βρίσκουν σύμφωνο, δηλαδή προβλήματα σε τράπεζες ορισμένων χωρών που λέτε. Δεν είναι κάτι που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε πολλά στοιχεία για κάτι τέτοιο. Πρέπει να προηγηθούν τα τεστ αντοχή, τα stress δηλαδή και αυτή η εξολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών. Ήδη τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουν κάνει πάρα πολλά οι τράπεζες για να ενισχύσουν τα αποθεματικά τους, να ενισχύσουν τους ισολογισμού τους. Εδώ μιλάμε για τα εναπομένοντα προβλήματα. Τώρα τι πρόβλημα μπορεί να προκύψει αυτό το πρόβλημα, το ενδεχόμενο θα αντιμετωπίζεται με βάση τις, ε, ε, τα, τις μεθόδους και τα μέτρα που περιέγραψε και δεν θα δίνεται μια λευκή επιταγή. Τώρα στην άλλη σας ερώτηση, οι χρηματοπιστωτικές αγορές, οι τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, θα υπάρχουν και κάποιοι κανόνες ε, κρατικοί που περιλαμβάνουν και ένα ανταλλάξει το ποσό bail-in όπως είπαμε. Μετά θα δούμε ε, μέχρι που φτάνουν αυτά τα κονδύλια της χώρας. Αν λοιπόν ξεπερνούν κατά πολύ τα προβλήματα και τα απαιτούμενα ποσά αυτά που μπορεί να διαθέσει μια χώρα, μετά θα μελετηθούν ε, ε, θα μελετηθούν τα ενδεχόμενα δυνατότητες για προσφυγή ε, στον μηχανισμό σταθερότητας. Αλλά είναι ε, στο τέλος της όλης αυτής διαδικασίας ε, η άμεση ανακεφαλαιοποίηση. Αυτό θα ήταν το τελευταίο, το τελευταίο βήμα. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να κάνω καμία εικασία αυτή τη στιγμή για το μέγεθος του προβλήματος. Εάν και εφόσον προκύψει. Αλλά σας λέω θα το αντιμετωπίσουμε αν προκύψει. Ο Πάμπλο τώρα, εκ μέρου ε, του ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω με βάση στοιχεία της Eurostat η Ευρωζώνη φαίνεται να βγει και από την ύφεση. Λέτε, σε κάποιες χώρες έχουμε σημαντική μείωση ε, του ε, δημόσιου ελλείμματος, βελτίωση επίσης ε, του ισοζυγίου πληρωμών. Όμως από το 1999 και μετά για ένα εξάμεινο πρώτη φορά που έχουμε εμπορικό πλεόνασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης βελτιώνονται οι εξαγωγές, ελέγχεται καλύτερα το χρέος από τις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είμαστε αισιόδοξοι με όλα αυτά. Όμως, η πίστοση που δίνεται και ιδίω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλο και μειώνεται. Και ένα από του λόγου που μα είπατε κι εσεί είναι ο κατακαιρματισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών και είπατε και συμφωνώ μαζί σα ότι η Τραπεζική Ένωση είναι μια λύση. Είναι όμω μια μακροπρόθεσμη λύση. Πολλέ και διάφορε ήταν οι αναγγελίε για σχέδια και πλάνα, αλλά λίγα από αυτά συγκεκριμενοποιήθηκαν. Εσείς είπατε ότι αυτό θα είναι προτεραιότητα για εσά και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι αν δεν υπάρχει πίστοση, αν μειώνεται η πίστοση, μειώνονται οι χορηγήσει, αυτή η τόσο ευκταία ε, ανάκαμψη δεν θα είναι εύκολα εφικτή. Και δεν υπάρχουν ε, σχέδια πολύ σαφή, πολύ συγκεκριμένα για τις ΜΜΕ. Τι μπορεί να κάνει έκτη και τι παραπάνω μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πρέπει να βάλουμε το ρολόι να τρέχει γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Άρα τι θα πει αυτό. Μπορώ να απαντήσω για όσο χρόνο θέλω. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Το κατά πόσο πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι όχι. Ναι, εγώ νομίζω ότι ναι, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Υπάρχουν λόγοι, βλέπουμε σε αρκετές χώρες και συνολικά στην Ευρωζώνη έχουμε πλέον εξέλθει από την ύφεση και σε κάποιες άλλες χώρες μπορούμε να έχουμε ενθαρρυντικά σημάδια, έχουμε μια αύξηση των θέσεων εργασίας, ανάκαμψη της οικονομίας, εύθραυστη, αλλά ε, λόγια ανησυχία, ε, συγγνώμη, υπάρχουν παρόλα αυτά. Τώρα, για τις ανησυχίες που εκφράσατε ως προς τις ΜΜΕ, πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα μπορεί να ανακάμπτει η οικονομία και μόλις ανακάμψει στις χώρες αυτές θα χρειαστεί ε, πίστοση για τις ε, ε, επιχειρήσεις και αν αυτό δεν μπορεί να δοθεί, αυτή η πίστοση δεν μπορεί να δοθεί, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν θέσεις εργασίας και να μειωθεί η ανάπτυξη. Η Τραπεζική Ένωση με πεπισμένος ότι είναι η δομική, η διαρθρωτική λύση για αυτό το ζήτημα και κάνω ό,τι μπορώ, πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε επιτύχει μεγάλη πρόοδο. Είπατε ότι είναι μακροπρόθεσμα αυτό το βράχι πρόθεσμο μέτρο είναι τα προγράμματα που έχουμε. Και είπατε εσείς ότι δεν αποδίδουν και καταλαβαίνω, καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Η κατάσταση αυτή είναι ως εξής. Έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κυρίως, οι οποίες υλοποιούνται. Η δυνατότητα της Τράπεζας Επενδύσεων να, να μπορεί να ε, δώσει κάποια βοήθεια έχει πλέον ε, ενισχυθεί ε, την άνοιξη και χρειάζονται και νέες πρωτοβουλίες. Είναι κατεπήγον αυτό και γι' αυτό το θέμα αυτό θα μπει και στο Eurogroup και στο ECOFIN το Σεπτέμβριο και θα μιλήσουμε με Κομισιόν, ΕΚΤΑ και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δούμε τι πρόοδο έχουν επιτελέσει με τι πρωτοβουλίε που έχουν αναλάβει ή θα αναλάβουν. Γιατί όπω είπατε, πάρα πολύ σημαντικό είναι η ροή των πιστώσεων, ε, οι χορηγίε προ ΜΜΕ να ε, επανέλθουν ε, σε κανονικού ρυθμού. Ο Βέρνερ τώρα. Ε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τις απαντήσεις του συνάδελφο Μπέλντερ σχετικά με την εξυγίανση τραπεζών. Πρέπει όμως να είμαστε πιο ειλικρινείς και αυτό ισχύει και για τους συναδέλφους. Ε, σε κάποιες χώρες χρειάζονται οπωσδήποτε μεταρρυθμίσεις. Πάει και τελείωσε. Πρέπει να δούμε και να πούμε πώς θα παρακολουθούμε ε, τις τράπεζες και πώς θα γίνεται η εξυγίανση. Ε, υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την πρόταση γιατί με την πρόταση και το πρόβλημα είναι με την Κομισιόν και την αρχή της το πρόβλημα της χειόδους τραπεζικής το παρουσίασε χθε ο Μπαρνιέ. Τι θα κάνουμε με τα ε, περιουσιακά στοιχεία, τα, στοιχεία του ενεργητικού στο, στη σκιώδη τραπεζική. Και το άλλο που είναι σημαντικό είναι να συζητήσουμε για τις φορολογικές οάσεις που προβλέπεται για το ε, ε, σύνοδο των G20. Ε, διάβασα τι δεν πάει καλά τώρα τελευταία. Και η χώρα σας, ε, κύριε Υπουργέ, είναι υπαριθμόν ένα φορολογική όαση. Δεν είναι οι Βερμούδες. Η Ολλανδία είναι φορολογική ένωση ε, και εις ό,τι αφορά τις άδειες ευρεσιτεχνιών. εκεί εξοικονομούν φόρους πολλούς. Μπορείτε αυτό να το ανεχθείτε μακροπρόθεσμα. Στο Λουξεμβούργο επίσης υπάρχει και ένα άλλο, ε, υπάρχει άλλο σύστημα σχετικά με την ε, ε μη φορολόγηση των ε, τόκων. Δηλαδή κάποιοι πλουτίζουν σε βάρος άλλων. Εδώ χρειάζεται ειλικρίνεια και ο κύριος Μπέλντερ είπε ότι στο δεύτερο γύρο θα πληρώσουμε δυο φορές η δέξια η οποία είναι Ολλανδο-Γάλλο-Λουξεμβουργική επιχείρηση, ε, έχει ε, μια τράπεζα 100 δις ευρώ ε, και βέβαια, όπως λέει η κυρία Βόρτμαν Κόλ, τα 100 αυτά δις που είναι προβληματικές καταθέσεις, πώς θα αντιμετωπιστούν κάποια στιγμή ε, έχουν ακουστεί και κριτικές φωνές στην Ευρωομάδα. Αλλά εδώ χρειάζεται μεγάλη ειλικρίνεια. Αυτή λείπει πολύ και τη χρειαζόμαστε επιγόντως Και για την, να πω κάτι για την Ολλανδία. Α, και να πείτε και για την Ολλανδία που είναι φορολογική οάση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκεν για την ερώτηση. Σχετικά με το θέμα της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, πάντα ήξερα ότι η ειλικρίνεια μας πάει πιο μακριά, κρατάει περισσότερο. Καμιά φορά αυτό που πρέπει να πούμε εμείς οι πολιτικοί ε, μπορεί να μην ακούγεται θετικό, καμιά φορά ο κόσμος και οι χρηματαγορές ε, δεν θέλουν να ακούν αυτά που τους λέμε, αλλά πρέπει να τα πούμε. Εγώ προσπαθώ, θα προσπαθώ να είμαι ειλικρινής για όλα αυτά που είπατε. Και κάτι άλλο που, για το οποίο έκανε και ο, ε, ε πρόσθετη ερώτηση ο κ. Λάμπερτ. Εγώ ως υπουργό Οικονομικών της Ολλανδίας πιστεύω ότι είναι για το συμφέρον όλων να έχουμε ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο και αποτελεσματικό. Και πρέπει στη φορολογική πολιτική να δουλέψουμε, να συνεργαστούμε περισσότερο. Ναι, οι διαφορές των φορολογικών πολιτικών μεταξύ των χωρών παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους ε, ενδιαφερόμενους και να δουν ποιο, είναι, ποιο είναι το πιο ευνοϊκό καθεστώς ω Ολλανδική κυβέρνηση απευθύναμε επιστολή πριν από λίγες μέρες στην Ολλανδική Βουλή. Ίσως ε, σας ενδιαφέρει να τη διαβάσετε. Και ε, αναφέρουμε πολλά από αυτά τα θέματα για τα οποία μας ασκείται κριτική. Με τρόπο επιθετικό, όχι αμυντικό. Οπότε θα αλλάξουν κάποια πράγματα στους Ολλανδικού κανονισμούς και στις νομοθεσίες και τις συμφωνίες μας με άλλες χώρες και ένας λόγος για τον οποίο έρχονται για φορολογικούς λόγους πολλές επιχειρήσεις στη χώρα μας είναι ότι έχουμε φορολογικές συμφωνίες σε όλο τον κόσμο. Θα τις αναπροσαρμόσουμε, θα τις ε, τροποποιήσουμε για να υπάρχει ρήτρα κατά της απάτης όλες τις συμφωνίες αυτές, να ε, μην υπάρχει φοροαποφυγή, δηλαδή να, μην, να υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν φόρο σε καμιά χώρα κλπ. Τώρα όμως μιλώ ως Ολλανδός υπουργό. Εμείς ε, το χειριζόμεθα το θέμα αυτό. Δεν αποφεύγουμε τη συζήτηση, είναι σημαντική η συζήτηση και πολλά έχουμε να κερδίσουμε σε όλη την Ευρώπη αν συνεργαστούμε για τα φορολογικά θέματα. Πολλές πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται τώρα, μιλήσατε για την ε, G20 αλλά και ο Πρωθυπουργό Κάμερον, ο Πρόεδρος Ολλάντ έχουν λάβει πρωτοβουλίες για να μπει σε ανώτατο επίπεδο το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και πολλά βήματα έχουν ήδη γίνει. Τώρα, ε, μάχη κατά της φοροδιαφυγής και της απάτης στις 14 Σεπτεμβρίου. Αυτό το θέμα είναι ήδη στην ατζέντα του ΕΚΟΦΗΝ. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τον Δεκέμβριο του 2012 ο κ. Φαραμπό είχε αναλάβει να προβλέψει ένα χάρτη πορείας, ένα φύλλο πορείας για να καλύψει τις ανεπάρκειες της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα οικονομικά εργαλεία. Και ετοίμασε και την έκθεση τίσεων του Ευρωκοινοβούλου για το θέμα αυτό, όπου θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε υπέρ της κοινωνικής διάστασης για να τονωθεί ε, κοινωνία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, να στηρίξουμε τι καταθέσει και να αντιμετωπιστεί η κρίση με τον δημοσιονομικό ε, πυλώνα και έναν πυλώνα επίση ε, για την νομισματική πολιτική, ώστε να λειτουργεί και η Ευρωζώνη πιο εύρυθμα, αλλά και το δημοκρατικό πυλώνα, ώστε να υπάρχει νομιμότητα και θεμητό στι ευρωπαϊκέ αποφάσει με τελευταίο επιστέγασμα την Τραπεζική Ένωση. Μιλήσαμε πολύ για την Τραπεζική Ένωση τελευταία, αλλά οι υπόλοιποι πυλώνε σήμερα δεν είναι και πρώτε τι προτεραιότητες ε, των ευρωπαϊκών συζητήσεων. Το μόνο που είδαμε να προκύπτει με... στην τελευταία περίοδο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτό που λέμε τη συμβασιοποίηση των οικονομικών πολιτικών όπως ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν έχει και πολύ να κάνει με την ε, κοινοτική μέθοδο όπως τη γνωρίζαμε. Η ερώτησή μου και επειδή ακούγονται πολλά ανησυχητικά για το φιλοπορίας ε, του Φανρομπόη και μπορεί και να ανακληθεί η χρήση του, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην ημερήσια διάταξη θα προβλέψετε αυτό το φιλοπορίας, ε, ποιο θα είναι το μέλλον της, τουλάχιστον άμεσα το μέλλον μάλλον του φιλοπορία. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ κύριο Χουάν Γκόκ για τις ερωτήσεις. Για το φίλο πορείας, όπως ξέρετε, το Eurogroup. Και οποτεδήποτε προκύπτουν τέτοια ζητήματα, για να προετοιμάσει τη συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συζητά το φύλλο πορεία και έχει υπάρξει στι ημερήσει διατάξει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το φύλλο αυτοπορία εδώ και κάτι πόσο καιρό. Όμω δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα των συμβάσεων, ούτε μπορώ εγώ να σα δώσω τα τελικά πορίσματα για αυτό το ζήτημα, το ζήτημα των συμβάσεων. Ούτε να σας πω τι θα συμπεράνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ω προ αυτά, Όλε αυτέ οι έννοιε θα πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω. Νομίζω συζητιούνται εδώ και κάμποσα χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να σα δώσω τα δικά μου πορίσματα, όμω έχετε μάλλον δίκιο. Διότι στο συνολικό πλαίσιο του φύλου πορεία υπάρχει μεταξύ των στοιχείων διαφορά ταχύτητα. Κάποιοι από του πυλώνε, κάποια από τα στοιχεία και τα σκέλη προχωρούν γρηγορότερα με την Τραπεζική Ένωση να σύρει το χορό ω πρώτη προτεραιότητα. καλύπτοντα κενά και ενώ υπάρχουν ακόμα οικονομικά εργαλεία που συζητιώνται και δεν έχουν υπερατωθεί. Από αυτήν λοιπόν την άποψη, στο Sixpack και στο Tupac διαθέτουμε καινούργια εργαλεία, καινούργια μέτρα τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν. Ζωτική σημασία είναι λοιπόν ενώ συζητούμε αν θα προκύψουν νέα εργαλεία, να φανούμε σοβαροί στην υλοποίηση αυτών που ήδη υπάρχουν. Τα έχουμε ήδη θεσπίσει, προβλέψει και συμφωνήσει. Η δική μου λοιπόν προτεραιότητα σε αυτή τη φάση θα ήταν να υλοποιηθούν, να αξιοποιηθούν τα συμπεφωνημένα εργαλεία, τα υπάρχοντα. Και μετά βλέπουμε αν χρειαζόμαστε και επιπλέον. Ευχαριστώ. Για το ΕΛΚ τώρα η κυρία Λούλιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, είπατε με ικανοποίηση, εάν καλά κατάλαβα, ότι οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Συμβούλιο. Έχω ε, κάπως, διότι αμέσως μετά την δημοσίευση αυτών των συστάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη κιόλας δηλαδή. Οι αντιδράσεις ήταν πολύ αρνητικές από την πλευρά των ε, πολιτικών των εθνικών κρατών και μάλιστα ε, των υψηλόπεθμών. Ο πρόεδρος Ολόγκ δεν ε, ενοχλήθηκε να κάνει σχόλια αρκετά έτσι απλά λέγοντας ότι δεν μπορούν οι Βρυξέλλες να υπαγορεύουν στα κάτι μέλη τι να κάνουν. Και στο Λουξεμβούργο όμως η υπουργοί μίλησαν για επιταγές των Βρυξελών και ότι οι συστάσεις που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν εκτός του σωστού δρόμου. ήταν εσφαλμένες. Λοιπόν, τελείως διαφορετικά τα θέτουν ε, οι πολιτικοί των Εθνικών Κρατών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γιατί υπάρχει αυτή η παράλληλη παρουσίαση του ίδιου θέματος. Υποκρισία είναι. Εμείς ε, την νομιμότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματο θέλουμε να προσπιστούμε. Δεν πρέπει λοιπόν και το Eurogroup να τη συζητήσει αυτή την διπλή όψη του ίδιου θέματος και να δει τι μπορεί να κάνει για το θέμα. Κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, τις τελευταίους ε, λάμψατε δια της διακριτικότητάς σας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό ε, δεν είναι ίσως αντικειμενική αποτίμηση. Εγώ δεν το βλέπω ούτε για πλεονέκτημα, ούτε για προτέρημα μέλλον, ούτε για ελάττωμα. Αλλά ποια είναι η λόγια αυτής της συμπεριφοράς. Διότι αντλήσατε κάποια διδάγματα από το βάπτισμα του, πυρό, πυρός που λάβατε με την κυπριακή κρίση. Κρίση δυσχερέστατη να τη χειριστεί κανείς με ιδιαίτερη βεβαίως δράση και επιρροή στο πολιτική διάσταση του θέματος. Κατηγορηθήκατε για δεξιότητες ως πρόεδρος του Eurogroup, νέος ναι, πρόεδρος του Eurogroup, για πολιτικές επιλογές άστοχες. Και επειδή εσείς βρεθήκατε να είστε πρόεδρος του Eurogroup, δεν θα πρέπει την διακριτική ευχαίρεια που δείξατε ότι διαθέτεται να την χρησιμοποιείτε για τι εσωτερικέ αποφάσει του Eurogroup καλύτερα. Οι συγκυρίε εδώ θα σα επέτρεπα να βελτιώσετε λίγο ε, τον τρόπο που εκτελείτε το ρόλο σα. Θα ήθελα λοιπόν να μα πείτε κάτι γι' αυτό. Γιατί υπήρξατε τόσο διακριτικό ω προ τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ευχαριστώ κυρία Λουλή για τις ερωτήσεις σας και ευχαριστώ για τη στήριξή σας για την ε, πολιτική μου, την, ε, τη, της παρουσίασής μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι θα παραμείνω παρόν ε, στην ευρωπαϊκή πολιτική και στο τι γίνεται στις Βρυξέλλες, προς εκεί που είμαι άποψη ενώ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δεν ε, προβάλαμε αρκετά το τι κάναμε και γιατί το κάναμε. Νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία ω υψηλόβαθμη πολιτική να μιλάμε για το τι κάνουμε. Διότι μόνο έτσι δείχνουμε πώ θέλουμε να αναχαιτήσουμε την κρίση, τι πρέπει να γίνει, πόσο σκληρή είναι η πραγματικότητα, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και το καθεξή. Σε ό,τι αφορά τι συζητήσει για τι αναχώρασει τάσει, Ναι, θα πρέπει να περάσουμε μετά από συζήτηση στο Eurogroup ομοφόνο οι συστάσει. Το ίδιο και στο ΕΚΟΦΗΝ. Και ναι, άκουσα τα σχόλια κάποιων από του εθνικού ε, πολιτικού, του πολιτικού των κρατών μελών. Νομίζω όμω, και πρέπει να σα το πω, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, και μετά βέβαια και το Συμβούλιο και το καθεξής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να ε, επιδώσει τις συστάσεις και να πει στις χώρες τι δεν πάει καλά στους τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τη μακροοικονομική αναδιάρθρωση, ανάταξη και τις μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το κάνει αυτό και είναι δική της αρμοδιότητα. Έπειτα οι χώρες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά με σοβαρό και αποτελεσματικό τρόπο. Πώς θα γίνει αυτό. Σας είπα το παράδειγμα του συνταξιδοτικού συστήματος. Εάν ένα συνταξιδοτικό σύστημα δεν έχει εξυγχρονιστεί ποτέ, εάν καθόλου δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τι μελλοντικέ προκλήσει, ε, χρειάζονται μεταρρυθμίσει. Ο τρόπο τώρα που θα γίνει αυτό είναι κάτι που το αποφασίζουν οι εθνικοί πολιτικοί. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι ο ορθό τρόπο να γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν λοιπόν επιταγέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Όλε οι διαδικασίε ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πράγματα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των αρχηγών και κυβερνήσεων. Εκείνοι αποφάσισαν ότι έτσι θα είναι η διαδικασία. Εκείνοι αποφάσισαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τι ε, διατυπώνει τι συστάσει. Τώρα θα πρέπει να τι πάρουν και σοβαρά υπόψη του όμω. Πώ θα το κάνουν αυτό. Διαφορετικέ μεταρρυθμίσει που χρειάζονται ε, και όλα τα υπόλοιπα είναι εθνικέ αρμοδιότητε. Εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα κάτι μελη τότε η Επιτροπή θα αξιολογεί και θα αποτιμά κατά πόσον έγινε με ορθό ή όχι τρόπο. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές αρμοδιότητες, διαφορετικές ευθύνες, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η σημασία του ρόλου της στην διατύπωση των συστάσεων είναι καθοριστική. Ευχαριστούμε. Έχουμε καθυστερήσει λίγο. Θα πρότεινα λοιπόν να ακούσουμε τις επόμενες δύο ερωτήσεις μαζί. Η κυρία Τουρούνεν και ο κύριος Σβάμπ θα μιλήσετε το ένας μετά τον άλλο η Έμιλη πρώτη και μετά ο Αντρέ. Και μετά οι υπόλοιποι τρει θα μιλήσετε και τρει ε, ένα μετά τον άλλο, αφού ακούσουμε τι απαντήσει στην Έμιλη και τον Αντρέ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, διότι έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Έμιλη. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ήθελα να επανέλθω σε κάποια από τα ζητήματα που θίξατε εσείς και οι μομιλητές μέχρι τώρα. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι τα νέα στοιχεία του ΑΕΠ, ότι βγαίνουμε σιγά-σιγά από την ύφεση, βγήκαμε από την ύφεση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε ε, συζητήσει το ενδεχόμενο ε, αντιμετώπισης ε, της, των μη επαρκών θέσεων εργασίας Επίση, ό,τι αφορά την αναθεώρηση των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών, πάρα πολλέ κριτικέ ακούστηκαν για, την, ε, για το εγχείρημα αυτό μέχρι τώρα ε, και η άσκηση παρακολούθησης και τα stress test και το τι έγινε μετά, εκτός της μεθόδου και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκε. Είπατε ότι δεν θα πρέπει να αμφιβάλλει κανείς γιατί το ότι είναι ποιοτικό το σύστημα αξιολόγησης των στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών και είπατε ότι θα γίνει από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Επειδή υπήρξαν όμως αυτές οι κριτικές, εσείς πώς ε, σκοπεύετε την ποιότητα αυτή να την διασφαλίσετε. Ευχαριστώ. Έχω λίγο χρόνο, λιγότερο από ό,τι είχε προβληθεί. Απαντήσατε στον κύριο Λάγκεν για την ε, απάτη και την φοροδιαφυγή. Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για ε, φορολογική πολιτική στις εταιρείε. Το κράτος μέλος όμως θα πρέπει να μην προσφέρει ευνοϊκή πολιτική. Μιλήσαμε πολύ για την Ελλάδα, δεν θέλω να προσθέσω πολλά. Πάντως το πρωταρχικό πλεόνασμα είναι βασική προϋπόθεση μετά από τις δημόσιες ανακοινώσεις για να αποφασιστεί η μετέπειτα βοήθεια. Το δημοσιονομικό αυτό πλεόνασμα, το πρωταρχικό δημοσιονομικό πλεόνασμα, τι σημαίνει για την απόφαση για τα επόμενα προγράμματα για την Ελλάδα. Τέλος, αφού έκανα μια σύντομη επίσκεψη με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς στην Ελλάδα, δεν θα ήταν καλό να... Ε, προσφερθεί αυτό το task force και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η Ελίζα Φερέιρα είπε ότι πολλές φορές είναι παραπλανητικά τα στοιχεία και αν υπάρχουν άνθρωποι επιτόπου που μπορεί να το ε, ε, βοηθήσουν να λυθεί αυτό το πράγμα τότε θα επιτευχθεί και μεγαλύτερη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Uh, thank you for your questions. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, σιγά σιγά βγαίνουμε από την ύφεση. Τώρα, Ανάπτυξη χωρίς απασχόληση, ο κίνδυνος αυτός. Σε κάποιες χώρες βλέπουμε ότι ξαναγυρίζει η ανάπτυξη, με μεγέθυνση και βελτιώνεται η οικονομία. Αυτό όμως παίρνει χρόνο μέχρι να ξαναβελτιωθεί η απασχόληση. Καμιά φορά ε, παρουσιάζεται ανάπτυξη, αλλά αυξάνεται παράλληλα για ένα διάστημα και η ανεργία. Στην αρχή μιας κρίσης ε, πέφτει η ανάπτυξη ενώ δεν ανεβαίνει αυτόματα ψηλά η ανεργία. Πάντα υπάρχει μια χρονική υστέρηση δηλαδή μεταξύ ανάπτυξης και απασχόλησης. Οπότε δεν με απασχολεί ε, θα υπάρξει μια χρονική υστέρηση μεταξύ της επανέναρξης της ανάπτυξης και μετά της ε, απασχόλησης. Ε, τώρα για τα stress test. Αυτό υπογραμμίζει την ε, ανάγκη να το κάνουμε σωστά αυτή τη φορά. Πώς θα το διασφαλίσουμε. Ε, βεβαίως είναι κυρίως ευθύνη της ΕΚΤ. Θα ζητήσουμε από την ΕΚΤ να μας ενημερώσει πώς θα οργανώσει τη διαδικασία αυτή και όπως τόνισα σήμερα θα συνεχίσω να τονίζω και όλοι ότι θα πρέπει να είναι διεξοδική διαδικασία πλήρη σε βάθος με ανεξαρτησία και για να γίνει σωστά και χρονικά πρέπει να συμμετέχουν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και ιδιωτικών επιχειρήσεων εταιριών. Ο κύριος ΣΒΑΠ μίλησε για την κοινή φορολογική πολιτική. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούν ότι αυτό είναι το καλύτερο. Να πάμε άμεσα σε κοινό επίπεδο πια φορολογικής πολιτικής, κοινή φορολογική ε, πολιτική. Νομίζω ότι πιο πρακτικό θα ήταν, δεδομένη της κατάστασης, να δούμε το συντονισμό, την κοινοποίηση πληροφοριών, ε, την εναρμόνιση, σταδιακά. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε άμεσα στην τελική φάση και να πάμε απευθείας να κάνουμε κοινή φορολογική πολιτική. Δεν μας βοηθήσει κάτι τέτοιο πολλά ωφέλη μπορούμε να αποκομίσουμε σταδιακά ε, και σιγά σιγά θα επιταχύνουμε στον ε, συντονισμό, την εναρμόνιση, την ε, κοινή ενημέρωση κλπ. Η έκτη είναι καλή εδώ. Τώρα για το Task Force, ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλες χώρες που δεν είναι μέσα σε προγράμματα και το κάνουμε. Υπάρχουν χώρες που στηρίζονται στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται με εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ, που πηγαίνουν σε πολλές χώρες επιτόπου για να βοηθήσουν. Ω ειδική ομάδα, task force. Ναι, η δυνατότητα υπάρχει και εφαρμόζεται ήδη, βεβαίω. Ωραία. Ρομπέρτο. Ρομπέρτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να σας ζητήσω να μας πείτε λίγο περισσότερα για αυτή την έθραυστη ε, ανάκαμψη. Πώς τη βλέπετε την ε, φύση της. Από πού προκύπτει αυτό. Επειδή η εκαθάριση του χρέους ε, λειτουργήσε αρκετά, επειδή παρά αυτήν την ε, καθάριση... δεν ε, μπόρεσε να υπάρξει και μετριασμό στην ταχύτητα τους τελευταίους μήνες περισσότερος χρόνος για τη Γαλλία χρέη της, ε, του δημόσιου τομέα στην Ιταλία και ούτω καθεξής. Όπως λοιπόν ορθώς λέτε τώρα, έχουμε ένα νέο ε, ισχυρό εργαλείο, το Tupac, και Πώς το βλέπετε εσείς αυτή τη σοβαρή ευθύνη να χρησιμοποιηθεί με σωστό τρόπο ώστε να μην υπάρξει επικάλυψη μεταξύ της ε, ανάπτυξης και της ε, ανάγκης για δημοσιονομική ισορροπία και των κοινωνικών αναγκών από την άλλη. Αυτό είναι ε, η επόμενη ερώτησή μου και επίσης πολύ γρήγορα Δεν πρέπει να υπάρχει και ένα δίχτυ ασφαλείας μετά την ε, έξοδο κάποιων χωρών από το πρόγραμμα της Τρόικας. Δεν θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα και για άλλες χώρες να μπορούν να κάνουν ε, χρήση των ορισματικών νομισματικών συναλλαγών. Ευχαριστούμε. πολύ κυρία ε, κύριε πρόεδρε ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση του κυρίου Σφαμπ την οποία δεν απαντήσατε και έχει να κάνει με το πρωτογενές πλεόνασμα που παρουσιάζει ήδη η Ελλάδα και το οποίο είναι και μεγαλύτερο αισθητά από το αναμενόμενο. Ε, ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η προϋπόθεση θα ξεκινήσει μια συζήτηση για ελάφρυνση του χρέους και των μέτρων ούτως ώστε να υπάρξουν αναπτυξιακές πνοές γιατί όπως ξέρετε συνθλίβεται η κοινωνία αλλά και η πραγματική οικονομία ε, και αυτό δεν είναι προς όφελος του τελικού στόχου. Και παράλληλα θέλω να ρωτήσω αν στο Eurogroup ασχολείστε με τα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων. Πρόσφατα απασχολεί πολύ τη χώρα μας μια α, ε, απέτηση από την Τρόικα να κλείσουν αυτόματα τρεις αμυντικές βιομηχανίες ενώ η άποψη του αρμόδιου Υπουργού, του Υπουργού Οικονομικών του κ. Στουρνάρα, είναι ότι θα ήταν μεγαλύτερο το όφελος αν διαρθρωθούν εν λειτουργία. Ε, ήθελα να ρωτήσω αυτό το θέμα επειδή απασχολεί πολύ τη χώρα μας είναι και είμαστε σε μια ευρεία πολιτική ιδιωτικοποίησεων αν απασχολεί και εσάς για να γίνουν οι καλύτερες να πάρθουν οι καλύτερες αποφάσεις προς όφελος της ίδιας της οικονομίας και των στόχων. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω τη σαφή σα δήλωση ότι η Ευρωομάδα θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να παραμείνει στο σωστό ρυθμό. Στην πράξη όμως αυτό μακροπρόθεσμα θα είναι αποτελεσματικό και λειτουργικό αν τα κράτη-μέλη θέσουν το κοινό καλό μπροστά από τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό δεν γίνεται παντού. Ακούσαμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος, οι Γερμανοί ε, δεν πείθονται πάντοτε γι' αυτό. Και την τελευταία εβδομάδα ακούσαμε ότι κάποιες συστάσεις της Κομισιόν ε, δεν γίνονται δεκτές. Πότε θα φτάσουμε πιστεύετε σε ένα στάδιο όπου θα είμαστε σίγουροι για την πρόοδο η οποία θεωρώ ότι ε, εξασφαλίζεται περισσότερο από τα μέτρα που προτείνει ο Μάριο Ντράγκη. Το Asset Quality Review Πώς θα είμαστε βέβαιοι ότι ε, θα οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα όχι μόνο μέσα στην ευρωζώνη αλλά και εκτός αυτής. Επίσης, για τις αδυναμίες των τραπεζών. Αν ο ESM ε, θα μπορεί να συμβάλλει στην ανακεφαλαιοποίηση, πώς θα είμαστε βέβαιοι ότι θα επαρκέσει για να ε, καλύψει τα προβλήματα των τραπεζών. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω αν τις ε, κατέγραψα όλες, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο γίνεται καλύτερα. Η πρώτη ερώτηση αφορά την τωρινή ανάκαμψη μετά την ύφεση, από πού προέρχεται, τι άλλο ε, χρειάζεται για να διατηρηθεί η ανάκαμψη. Νομίζω ότι προέρχεται από σειρά μέτρων η ανάκαμψη αυτή και η ό,τι αφορά την ε, εξυγένση τραπεζών, τις μεταρρυθμίσεις στον δημοσιονομικό τομέα και δράσεις που ανέλαβε η ΕΚΤ βέβαια, ε, ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στην Ευρωομάδα και την οικονομία της. Τώρα, πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Πρέπει να φροντίσουμε να μην σταματήσουμε εδώ εις ό,τι αφορά τις ε, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, γιατί όπως είπα πολλά πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή τους. Ε, είναι σημαντικό επίσης ε, να κρατήσουμε έναν ε, ρυθμό ε, σωστό στη λήψη μέτρων για τα ελλείμματα και είναι σημαντικό να δουλέψουμε, όπως σας είπα, και για την Τραπεζική Ένωση. Έτσι λοιπόν, πρόκειται κυρίως για εμπιστοσύνη, θα πρέπει ο δημοσιονομικός τομέας να ξαναλειτουργήσει σωστά και να κάνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και στον έξω, έξω κόσμο. Τώρα, ε, για την ε, Ιρλανδία ε, θα υπάρξει βοήθεια για να ξαναμπεί σταδιακά στις χρηματαγορές. Πήγε καλά το πρόγραμμα της Ιρλανδίας και θα βγει από το πρόγραμμα η χώρα αυτή αλλά θα υπάρξουν υποστηρικτικά μέτρα για να ε, υπάρξει σταδιακή έξοδος. Δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες, γιατί αυτό ρωτήσατε τι θα κάνουμε συγκεκριμένα, ποια θα είναι η υποστήριξη συγκεκριμένα. Πάντως θα υπάρξει υποστήριξη, αυτό μπορώ να σας πω, για να είμαστε βέβαιοι ότι θα βγει σωστά στις αγορές και μόνιμα, όχι για λίγο μόνο. Ε, άλλη ερώτηση δεν έχω. Α, η κυρία Κράτσα για την Ελλάδα μας, μας, ρώτησε. Η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλά σε πολύ δύσκολη εποχή για να επιτύχει στον προϋπολογισμό πρωτογενές ε, πλεόνασμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, ήταν μία από τις κέρυες προϋποθέσεις. Τώρα, για τα πρόσθετα μέτρα. Τα πρόσθετα μέτρα θα μπορούσε να είναι ελάφρυνση του χρέους ή ένα άλλο που συμφωνήσαμε και να πω πρώτα ότι θα αξιολογήσω με το που βρισκόμαστε στο πρόγραμμα και σε σχέση με τη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό θα γίνει τον Απρίλιο του χρόνου και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κι άλλα υπό τον όρο ότι θα, πληρεί, θα πληρώσει όλους τους όρους του προγράμματος η Ελλάδα. Κάποια μέτρα αναφέρθηκαν που ενδεχομένως θα εξεταστούν για τη βιωσιμότητα του χρέους αν χρειαστεί. Το ένα είναι περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στα διμερή δάνεια το άλλο είναι περαιτέρω ε, αλλαγή της συγχρηματοδότησης για να έχει καλύτερη πρόσβαση η Ελλάδα στα διαρθρωτικά ταμεία. Δεν θέλω να κάνω εικασίες ε, ούτε για το πού θα είμαστε τον Απρίλιο σε σχέση με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους ή το τι μέσα και μηχανισμοί θα χρειαστούν επιπροσθέτως. Η ιδιωτικοποίηση είναι μια διαδικασία η οποία δεν πηγαίνει τόσο γρήγορα και τόσο καλά όσο ελπίζαμε και όσο ήλπιζε η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα για το αν θα το ξανασκεφτούμε, αν θα γίνει αναδιάρθρωση, μπορεί να γίνει συνδυασμό των δύο. Η ιδιωτικοποίηση όμως είναι επίσης απαραίτητη για την οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος. Είναι ένα από τα στοιχεία που θα συμβάλλουν και στη βιωσιμότητα του χρέους. Οπότε η αναδιάρθρωση από οικονομικής άποψης ε, ε, μπορεί να είναι απαραίτητη, αλλά δεν συμβάλλει στο πρόγραμμα και εμείς πρέπει να τηρήσουμε τους στόχους του προγράμματος. Ο κύριος Βολφ είπε ότι πρέπει να παραμείνει ακέραιη η ευρωομάδα. Αυτό θα πρέπει να γίνει βάζοντας το κοινό καλό ε, πάνω από τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό το έγραψα. Μου άρεσε πολύ αυτό που είπατε. Το κοινό καλό πάνω από τα εθνικά συμφέροντα. Και πότε θα είμαστε ασφαλείς ρωτάτε. Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί βεβαίως. Αλλά μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν με τη συνεργασία, βάζοντας πάνω από όλα το κοινό καλό, τηρώντας όλες τις συμφωνίες για τις μεταρρυθμίσεις, διαφορετικές στην ε, Τραπεζική Ένωση, δημοσιονομικές συμφωνίες, να κάνουμε ό,τι αποφασίσαμε και συμφωνήσαμε. Είναι καλό και για την εμπιστοσύνη. Τώρα για τις τράπεζες εκτός ευρωομάδας. Η Τραπεζική Ένωση, όπως είπα, είναι θέμα του ΕΚΟΦΗΝ. Γιατί, διότι εξορισμού ε, δεν αφορά την Ευρωζώνη και εξέφρασα την ελπίδα και άλλες χώρες που δεν είναι στην Ευρωομάδα να μπουν στην Τραπεζική Ένωση και να μπουν στον SSM, δηλαδή να είναι επίσης ε, μέρος του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης. Αλλά κατά τα άλλα η Τραπεζική Ένωση θα συμβάλλει στην εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ τραπεζών μέσα και έξω από την Ευρωομάδα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και για το ότι μείνατε λίγο παραπάνω ώστε να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Φυσικά θα δούμε πιθανές ημερομηνίε ώστε να προσκαλέσουμε το 2014 και βέβαια εφόσον προκύψει κάτι επίγον θα σας ε, ξανακαλέσουμε. Ελπίζω να μην χρειαστεί βέβαια, αλλά είμαι βέβαια ότι θα έλθετε σε περίπτωση που σας ε, απευθύνουμε πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Την ε, Προεδρία θα την αναλάβει για λίγο αντιπρόεδρος. Έχω κάποιες ε, πήγουσες ε, υποχρεώσεις. Θα επανέλθω για τις ψηφοφορίες. Good morning everyone. So we move to the... Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Περνάμε στο σημείο 4. Ο Αντιπρόεδρος Στόλογιαν, ο εισηγητής, του δίνω το λόγο. Uh, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να συζητήσουμε τις τροπολογίες στην έκθεσή μου. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι αυτή η έκθεση αναφέρεται στο πρόγραμμα της Ένωσης 58 εκατομμύριων ευρώ για την περίοδο 2014-2020 για τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος για τα Διεθνή ε, Πρότυπα Χρηματονομικής Πληροφόρησης, το Ταμείο Εποπτείας με στόχο και, την, ε, και τα λογιστικά πρότυπα και το Συμβουλευτικό Σώμα με στόχο την έγκριση των λογιστικών πρότυπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο εργαζόμουν για αυτή την έκθεση, συναντήθηκα μαζί με τους κοιόδης ηγητές, αλλά και με ακαδημαϊκούς και επαγγελματίε από τους εθνικούς ε, και διεθνείς τομείς ε, των ληστικών προτύπων. Συναντήθηκα επίσης και με επαγγελματίε που χρησιμοποιούν αυτά τα πρότυπα. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στις συζητήσεις. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό, για να μην ανησυχείτε, ότι τα ξεκαθαρίσαμε και όλα. Γιατί δεν τα ξεκαθαρίσαμε όλα, διότι υπάρχουν διαφορές, διαφωνίες μεταξύ ακαδημαϊκών επαγγελματιών και αυτών που καθορίζουν τα πρότυπα για το ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Η ΕΚΟΝ ζητήθηκε λοιπόν, από την ΕΚΟΝ μάλλον, να αναβάλει την ψήφιση αυτής της έκθεσης για δύο λόγους. Κανονικά θα ψηφίσταν σήμερα. Ποιοι είναι οι λόγοι. Πρώτον, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να καταλήξουμε σε καλέ συμβαστικέ τροπολογίε διότι θέλουμε να έχουμε μια πάρα πολύ ισχυρή πλειοψηφία που θα στηρίξει αυτή την έκθεση. 78 μόνο είναι οι τροπολογίες στην έκθεση αυτή. Όμως, τα ζητήματα που θέτουν είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της λογιστικής και των λογιστικών προτύπων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεύτερος λόγος. Την εβδομάδα αυτή αναμένουμε τις προκαταρκτικές συστάσεις ε, του ειδικού συμβούλου κ. Μάιστατ στον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της ε, διαδικασίας έγκρισης ε, στα κράτη-μέλη. Τι σημαίνει αυτό, ότι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες ε, συγκεκριμένες ε, ε, εξελίξεις και συγκεκριμένα αιτήματα. Η Κομισιόν θα ήθελα αυτή την εβδομάδα να μας ε, κοινοποιήσει αυτές τις προκαταρκτικές συστάσεις. Τι είναι πιο βασικό στην όλη συζήτηση. Ουσιαστικά ότι αυτό είναι η αρχή μόνο. Του χρόνου, με βάση τη δουλειά ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ολοκληρώσει την του αντικτύπου των 8 χρόνων από τη χρήση του IFRS, αυτού του συστήματος δηλαδή για την ε, χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα χρησιμοποιηθεί και για την ε, αναθεώρηση και του, των διεθνολογιστικών προτύπων. Για να έχουμε λοιπόν καλές συμβαστικές τροπολογίες, θα πρέπει τις ε, τροπολογίες μας ε, να τις ε, κρίνουμε με βάση κάποια συγκεκριμένα θεμελιώδη στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, η οικοχρηματοοικονομική πληροφόρηση, αν έχει καλή ποιότητα, αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό για τις οικονομικές αγορές. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο της οικονομικής διακυβέρνησης. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο οικονομικό κόσμο χρειαζόμαστε μία ενιαία δέσμη προτύπων, λογιστικών προτύπων και προτύπων ελέγχου. Άρα θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση των διαφορετικών προτύπων που ισχύουν στον κόσμο. Αυτό είναι ένα στόχος που τον επανέλαβε και η ομάδα των 20. Εφαρμόζονται βέβαια αυτά τα πρότυπα σε πάνω από 100 δικαιοδοσίες, αλλά αν δεν τις δεχτούν ε, οι ΙΠΑ δεν πρόκειται να έχουν αποτέλεσμα. Όλο και περισσότερες δικαιοθεσίες δέχονται ότι η πρώτη ρύθμιση ε, είναι καλύτερο να γίνει από έναν εξάρτητο ε, φορέα που θα προβλέπει τις σωστές διαδικασίες για μια διαδικασία ε, που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και ε, λογοδοσία. Αυτοί οι ανεξάρτητοι φορείς θα πρέπει βέβαια να εργάζονται προς το κοινό καλό, προς το κοινό συμφέρον. Η διαδικασία δε κατάρτισης των προτύπων αυτών στη Εθνική θα πρέπει να είναι συνεργατική, δηλαδή να συμμετέχουν όλοι και η Εθνική ε, Αρμοδιφόρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν μηχανισμό έγκριση που ουσιαστικά την τελευταία, την ε, οριστική απόφαση την αφήνει στα χέρια της Ένωσης για τα πρότυπα αυτά. Αν ε, βέβαια υπάρχει ισχύ ότι αυτά, αυτή η διαδικασία είναι αποτελεσματική. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ε, εξίσου σημαντικό με τον καθαρισμό του προτύπου, είναι και η εφαρμογή του προτύπου. Αλλά η εφαρμογή του προτύπου είναι εφαρμογή και των ελεγκτών και των λογιστών. Τώρα έρχομαι στις τροπολογίες. Το σημαντικότερο θέμα που θίγουν οι τροπολογίες αυτές, μάλλον τα σημαντικότερα θέματα είναι τα εξή. Οι ευρωπαϊκές ε, ιδέες ε, της λογιστικής prudence, true and fair, stewardship, αυτές οι τρεις αρχές δεν είναι πλέον στο ενολικό πλαίσιο του ERCB. Αυτό είναι η πρώτη ανησυχία. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που προτείνουν αυτοί οι έννοιες να ενταχθούν στο ενοιολογικό πλαίσιο και στα λογιστικά πρότυπα και ζητούν επικαιροποίηση και για τους φορείς που ρυθμίζουν και καταρτίζουν τα πρότυπα. Υπάρχουν ανησυχίες πράγματι, όμως οι τροπολογίες δεν συνάδουν με την αρχή της ανεξαρτησίας αυτών που ορίζουν τα πρότυπα σε αυτό πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Όπως προείπα, γίνονται έντονες συζητήσεις για το θέμα αυτό επί του παρόντος. Επομένως, οι συμβιβαστικές τροπολογίες έχουν ως στόχο να διατηρηθεί η αρχή της ανεξαρτησίας και να γίνει επανεξέταση του θέματος βάσει της πρότασης της Κομισιόν η οποία ζητεί ε, μία μελέτη για να υπάρξει ανάθεση διαγωνισμού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονε οι οποίοι θα αναλύσουν τον αντίκτυπο των 8 ετών χρήση αυτών των προτύπων IFRS στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα πρέπει να γίνει, κατά την άποψή μα, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2014. Δεύτερη ανησυχία αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας έγκρισης. Και για το νέο ενεργητικό ρόλο του ΙΦΡΑΚ σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των προτύπων. Με βάση κάποιους όρους εργασίας που έχουν οριστεί από την Κομισιόν και με βάση το χρωματοδοτικό πρόγραμμα 2010-2013, πρόγραμμα που εγκρίθηκε από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Αυτές οι τροπολογίες έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και τη λογοδοσία. Αλλά και να σχετίσουν τη χρηματοδότηση με την υλοποίηση αυτών των προτάσεων. Οι συμβαστικές τροπολογίε έχουν ως στόχο τη διατήρηση ανεξαρτησία τη τεχνική ομάδα του ΕΦΡΑΚ. που έχει την ευθύνη να αξιολογεί τη συνεκτικότητα του IFRS με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Με βάση την πρόταση της Κομισιόν. Εμείς πιστεύουμε ότι μέχρι τα τέλη του Μαρτίου 2014 θα πρέπει να είναι έτοιμη αυτή η πρόταση. Και στις δύο περιπτώσεις, εάν το Ίδρυμα ΙΑΦΡΕΣ και το ΕΦΡΑΚ δεν υλοποιήσουν την πρόταση της Κομισιόν με βάση τις ε, αναθεωρήσεις αυτές, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, θα τεθεί θέμα αναστολή σημείωσης της χρηματοδότησης. Τρίτη ιδέα που προτείνεται μέσα των τροπολογιών είναι να περάσουμε σε αιτήσια έγκριση από Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη χρηματοδότηση των οργανισμών αυτών. Και συγκεκριμένα ότι δεν θα πρέπει να δώσουμε εξουσιοδότηση λευκό για 7 χρόνια σε αυτούς τους οργανισμούς. Η προτινόμενη σημαστική τροπολογία διατηρεί την πρόταση Κομισιόν για την ετήσια, αυτή, ε, τον ετήσιο έλεγχο μεταξύ δικαιούχων και Κομισιόν, αλλά εισάγει και το θέμα της ετήσιας αξιολόγησης της κομισιόν σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος, του προγράμματος ή των προγραμμάτων εργασίας και των μέτρων που προέρχονται από την ανάλυση που θα γίνει και από τους ανεξάρτητους εμπειρό Δηλαδή για δύο αναθεωρήσεις μιλάμε. Στην ουσία πρέπει να γίνει μέχρι τα τέλη Οκτώβρη 2014 για το FRS, τα Διεθνή Πρωτόκολλα οικονομική δηλαδή, Πληροφόρηση, Διακυβέρνηση και τις έννοιες, τα κόνσεπτ της λογιστικής και άλλη μία αναθεώρηση μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2014 για τα ζητήματα που σχετίζονται με το ΕΦΡΑΚ. Την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο οι εισηγητές, ε, ο εισηγητής μάλλον και οι σκιώδεις να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τις ε, σημαστικές μας τροπολογίες ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 23 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ Τεοντόρ για τους σοσιαλιστές. Ο κύριος Αλκαραούι. Σκιώδης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή που ήταν σχετικά σύντομος. Είναι πολύ καλό ότι λάβατε υπόψη την ε, πρότασή μας να αναβάλλετε την ψηφοφορία για να έχουμε καλύτερες συμβιβαστικές λύσεις και τονίσατε κι εσείς ότι ε, έτσι θα λάβουμε υπόψη μας και την ενδιάμεση έκθεση που τα εξετάζει αυτά και μπορεί το έγγραφο αυτό να περιέχει και πολλές χρήσιμες προτάσεις. Την επόμενη εβδομάδα στις συζητήσει μα θα τα λάβουμε υπόψη μα αυτά. Επί της ουσίας δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς για την συγχρηματοδότηση των ε, οργανισμών αυτών. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ξεκάθαρο το σύστημα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Αλλά θα πρέπει τα πρότυπα που θα αναπτυχθούν να είναι σύμφωνα και να συνάδουν με όλους τους κανόνες και κανονισμούς της Ένωσης. Και αν δείτε τις λογιστικές αρχές, πρέπει και αυτές να λαμβάνονται υπόψη στη δουλειά που γίνεται. Αν δεν γίνει αυτό σε επαρκή βαθμό, τότε θα είναι δύσκολο να συνεχιστεί η χρηματοδότηση στο επίπεδο που παρήχεται μέχρι τώρα και που παρέχεται τώρα. Ένα βασικό ζήτημα είναι ότι πολλοί από αυτή την εργασία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάμε για λογιστικά πρότυπα. Το 43% ε, των κονδυλίων προέρχονται από την Ένωση. Το γενικό συμφέρον πάντοτε πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Και εδώ, εις ό,τι αφορά την διαφάνεια και τις εγγυήσεις, νομίζω ότι πρέπει να τα παρακολουθούμε καλύτερα αυτά. Συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή λοιπόν να μην δώσουμε λευκό επιταγή για όλη την εξαετή περίοδο αλλά να τα παρακολουθούμε αυτά κάθε χρόνο και να βλέπουμε ε, τι ανάγκες υπάρχουν ούτως ώστε να είναι πιο ξεκάθαρη εικόνα μας για τα πράγματα σε αιτήσια βάση. Ε, νομίζω ότι θα προχωρήσουμε εδώ και περιμένω να το συζητήσουμε και άλλη φορά αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα Άλντε, ο κύριος Κλίντς, εισηγητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χτες με τον εισηγητή και τους Σκιώδης κάναμε μια συνάντηση και κάναμε κάποιες διαπιστώσεις. Καταρχήν σε μεγάλο βαθμό πέρα από πολιτικά όρια υπάρχει και ομάδες υπάρχει συμφωνία ότι, γιατί και θα το είδατε ότι ε, υποστηρίχθηκαν και κατετέθησαν από κοινού τροπολογίες από πολλές πολιτικές ομάδες. Ε, δεν μπορούμε να δώσουμε τελικά νούμερα εις ό,τι αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα χρειαστεί για την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων που πρέπει να υποστηριχθούν, όπως είπε και ο προλαλής σας. Είναι αυτονόητο αυτό και μας ενδιαφέρει όλους. Μας ενδιαφέρει να... Ε, συνεχιστεί η εξέλιξη των ε, αγορών. Ε, σημαντική είναι η σύνθεση του Συμβουλίου ε, και σημαντικό είναι πώς θα αναπτυχθούν τα πρότυπα γιατί θέλουμε οι λεπτομέρειες που διέκριναν το σύστημά μας στο παρελθόν θα εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη στα λογιστικά μας, ε, στο λογιστικό μας σύστημα. Εγώ έχω σχετικά καταθέσει τις τροπολογίες 38 και 42. Το συμβουλευτικό ρόλο του κ. Μάριστα δεν τον υποβαθμίζω και μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε και να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται τις προτάσεις τους. Αλλά να είναι απόλυτα σαφές ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, από ό,τι καταλαβαίνω, ε, θα ε, λάβουν ε, υπόψη πρώτα τις προτάσεις τις δικές τους. Επίσης νομίζω ότι οι προτάσεις θα πρέπει να έρθουν στο τραπέζι νωρίτερα από το Μάρτιο του χρόνου. αυτό ισχύει και για την τροποποίηση του κανονισμού 1606. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ είπε ότι χρειάστηκε ένας χρόνος για να τροποποιηθεί ε, ο κανονισμός και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε και ακόμη ένα χρόνο. Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι βέβαιο και συμφωνούν οι περισσότεροι συνάδελφοι, είμαι βέβαιος, ότι ε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το μέσο που έχουμε για να επηρεάσουμε τη δουλειά του Συμβουλίου στο βαθμό που είμαστε συγχρηματοδότες. Ε, αυτό πρέπει να είναι σαφές. Δεν θα ε, εκδώσουμε βέβαια, όπως είπα, εν λευκό επιταγή, επιταγή μέχρι το 2020. Θα πρέπει για να κρίνουμε την επόμενη δόση να δούμε πόσα θα είναι τα συνολικά κονδύλια που θα χρειαστούν και από πού θα δοθούν. Ο ιδιωτικός τομέας ε, και οι μεγάλες οργανώσεις ε, ε, ορκωτών λογιστών που θα συμβάλλουν και σε ποιο βαθμό θα χρηματοδοτήσουμε εμείς. Εκεί λείπουν ακόμα πληροφορίες. Ευχαριστώ κύριε Κλίντς. Ο κύριος Γκίγκολντ από την πλευρά των Πρασίνων. Επειδή αργούμε, δεν θέλω να επαναλάβω όλα τα επιχειρήματα εμείς δουλεύουμε και με τον εισηγητή και με τους σκιώδεις. Πιστεύω και εγώ ότι λόγω των σημαντικών ερωτήσεων που ετέθησαν εδώ στην ε, Επιτροπή και από τους εμπειρογνώμονες επίσης, δεν πρέπει να επιβεβαιώσουμε την ε, ισχύουσα δομή αμέσως θέτω ένα κέριο ερώτημα. Εδώ δεν πρόκειται μόνο για την ανεξαρτησία των οργανισμών που καθορίζουν τα πρότυπα. Ακόμα και αν έχουμε ανεξάρτητο παράγοντα, ε, το ερώτημα είναι υπάρχει ισορροπία και εκεί υπάρχει πρόβλημα με την τωρινή δομή. Αυτό ισχύει και για το, την ε, σόχα την, ε, και για το Συμβούλιο των Προτύπων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τα δούμε αυτά. Μην λέμε δηλαδή ότι μπορεί να συνεχίσει το σύστημα και είναι ανεξάρτητο. Ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται στις ε, ε, ε, λογιστικές ανάγκες και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά δεν ανταποκρίνονται και στην ανάγκη διαφάνειας που χρειάζονται το, ο κόσμος, χρειάζεται ο κόσμος και οι επενδυτές. Ευχαριστώ που είσαστε και σύντομος. Τέλος, ο κύριος Καμάλα για την ECR. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρω. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Στολόγιαν και τους άλλους ε, εισηγητές. Είναι σημαντικό το θέμα της συνεργασίας, δεν είναι πολιτικό το θέμα. Θέλουμε αυτό το δύσκολο θέμα των λογιστικών προτύπων να το αντιμετωπίσουμε πολύ καλά. Τώρα, κάποιες παρατηρήσεις, ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ακόμα μας ανησυχεί το αν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου και του ε, Ιδρύματος Λογιστικών Προτύπων ή ε, ε, προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. ανεξαρτησία δεν αρκεί για να διασφαλίσουμε ότι συνάδει με το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο το Ίδρυμα για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά. Επίσης, το θέμα της ενημέρωσης ε, είναι σημαντικό. Ε, Δεν ε, υπάρχουν στοιχεία σχετικά ε, μεταλογιστικά. Ε, ε, αναφέρεται ότι τα διεθνή πρότυπα δεν συνέβαλαν στην κρίση ενώ πολλοί χρηματοπιστωτικοί και τραπεζικοί οργανισμοί αναφέρουν το αντίθετο. Εδώ πρέπει να σταθμίσουμε τα πάντα πριν αποφανθούμε εμείς. Δεν είμαστε κατά των παγκόσμιων προτύπων. Δεν είναι καθ' αυτό κακή ιδέα. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε να μην παραγνωρίσουμε θέματα όπως stewardship, σύνεση, δικαιοσύνη, πραγματικο... ειλικρίνεια. Αυτά είναι αρχές που δεν πρέπει να παραμερίσουμε γιατί πολλές φορές ε, είδαμε ότι αυτά τα πρότυπα συνέβαλαν στην κρίση. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα. Ε, βεβαίως δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη χρηματοδότηση, αλλά θα πρέπει να βρούμε μια συμβιβαστική λύση όπως την προσωρινή χρηματοδότηση, μέχρι να βεβαιωθούμε και να πούμε ότι είμαστε με τη μία ή την άλλη άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έδωσα όμως το λόγο σαν πρόσωπο της ΓΚΟΕ και ζητώ συγγνώμη. Κύριε Κλούτε, έχετε το λόγο. Λόγω χρόνου δεν θα κάνω άλλα σχόλια. Ε, έχουν αναφερθεί πολλά από αυτά που εγώ είπα. Δεν θα σχολιάσω. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κλούτε. Άρα να δώσω εγκατακλείδη το λόγο στον εισηγητή κύριο Στόλογιαν. Στόλογιαν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά, όμως ε, αυτό το οποίο θέλω να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να μας πει αν είναι δυνατόν πότε μπορούμε να λάβουμε αυτές τις προκαταρκτικές συστάσεις του Ειδικού Συμβούλου. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομος, κύριε. Εκπρόσωπος Κομισιόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι στα γαλλικά η έκθεση και ολοκληρώνω το που να είναι η μετάφρασή της στα αγγλικά. Είναι θέμα ορών ουσιαστικά, ε, μέχρι να αντιλάβετε. Απλά δεν εξαρτάται από μένα Απολύτως, αλλά θα φροντίσω για την επόμενη εβδομάδα θα έχετε στα χέρια σας αυτό το έγγραφο. Κύριο Στόλογιαν, ε, σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές και θα ήθελα να απευθύνω ένα θέρμο ευχαριστώ στους κοιόδης για τις προσπάθειες που κατέβαλαν ώστε να έχουν συνομιλίες με πολλούς εκπροσώπους ε, ε, από, από τον τομέα αυτό ε, της ε, χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των λογιστικών ελέγχων. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Στόλογια. Θέλω να σας υπενθυμίσω απλά ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας ε, θα λάβει χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ημερομηνία για την ψηφοφορία. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη μερίσιας διάταξη, στο σημείο 5, που είναι η εξέταση των τροπολογιών σε το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οικονομικό έτος 2014. Η μα μας, ο κύριος Σβέν Γκίγκολτ, που εξαφανίστηκε. Α, έρχεται, εντάξει. Όσο τον περιμένουμε να πω ότι θα δώσουμε το λόγο μας στον κύριο Σβέν Γκίγκουλ, το οποίο είναι για αυτή την έκθεση. Well, suddenly uh, it's uh, all, quick here. Πολύ γρήγορα γίνονται όλα ξαφνικά, αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο θα εστιάσω στα σημαντικότερα και σε αυτά που δεν έχουμε ακόμη συζητήσει. Και επομένως θα εστιάσω και μόνο στα ποσά Νομίζω ότι έχουμε ξανασυζητήσει και έχουμε επιβεβαιώσει τις διαφορές μας για το κατά πόσο χρειάζεται μεγαλύτερο προπολογισμό η Ευρωζώνη, για το κατά πόσο χρειάζεται μεγαλύτερο περιορισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο ερώτημα είναι εάν απαντήσουμε καταφατικά στο πρώτο, αν θα πρέπει να υπάρχουν περικοπές στους τομείς οι οποίοι δεν συμβάλλουν τόσο πολύ στους στόχους της ε, Ευρώπης 2020 και αν χρειάζεται ε, αντίθετα να κάνουμε αυξήσεις ε, στους τομείς που ε, συμβάλλουν. Υπάρχουν πάλι συνήθεις διαφορές για το κατά πόσο θα πρέπει η αντικυκλική δαπάνη να έχει ένα πιο ε, ισχυρό ρόλο. Νομίζω ότι θα είναι κρίσιμες κάποιες ψηφοφορίες για αυτά τα ζητήματα, οπότε οι πλειοψηφίες θα έχουν το λόγο να αποφασίσουν. Όπως γνωρίζουμε, για τη διατύπωση ουσιαστικά έχουμε συμφωνήσει. Ό,τι αφορά τα ποσά και τις τρεις ΕΣΑ και την Eurostat ε, τις επισκέφθηκα. Και μου επιβεβαιώθησαν ότι οι ευρωπαϊκές αποπτικές αρχές χρειάζονται περισσότερους πόρους για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρα στην πολύ σημαντική τους δουλειά που εμείς τους αναθέσαμε με την νομοθεσία μας μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων. Υπήρξαν περικοπές ε, από την Κομισιόν ήδη, ε, μεγάλες περικοπές σε αυτά που είχαν προτείνει και ε, οι περικοπές αυτές ενισχύονται, γίνονται μεγαλύτερες με την πρόταση του Συμβουλίου. Και στην συνάντηση έγινε συζήτηση για το ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στα ποσά που έδωσαν οι ESA. Τώρα, σε ό,τι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα, από τον κύριο Νταμάχα μάθαμε ότι δεν υπάρχουν επαρκή σπόροι, υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσον ε, θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν. Είχα ζητήσει κάποια πόσα μπορούμε να τα ξαναπροτείνουμε, αλλά θέλω να θυμίσω στη Eurostat ότι αυτό βέβαια θα πρέπει να σημαίνει ότι πρέπει να το εφαρμόσουν το πρόγραμμα και όχι να διαλέξουν τι τους αρέσει και να μην ε, πραγματοποιήσουν ε, ό,τι δεν τους αρέσει, να μην εφαρμόσουν ό,τι δεν τους αρέσει. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε ως ένα βαθμό και το θέμα του ε, ποιες θα είναι οι άλλες, ποιες θα είναι οι άλλοι εκτελεστικοί οργανισμοί που θα δοθούν πόρους. Είχαμε προτείνει κάποιες περικοπές, αλλά μετά τη συνεδρίες των σχεδόν, οι περικοπές ε, γίνανε μεταφορά του κονδυλίου στο αποθεματικό στις περισσότερες περιπτώσεις. Εγώ λέω όμως για τα πρότυπα στον τομέα της χρηματοοικονομικής ε, πληροφόρησης και του λογιστικού ελέγχου να μπουν ε, στο αποθεματικό. Συζητήσαμε για το SB και το ΕΦΡΑΚ. Εγώ λέω να μπουν τα χρήματα στο αποθεματικό και σε ό,τι αφορά ε, την επικοινωνία για την Οικονομική Ονοσματική Ένωση. Αυτό το λέω γιατί θεωρήσαμε ότι ένα μέρος του παραγόμενου υλικού δεν ανταποκρίνεται ή δεν απαντά μάλλον ε, στα πολύ σημαντικά και πολύ κρίσιμα ερωτήματα που έχουν οι πολίτες μας και δεν είναι και πιστικά τα όσα γράφονται. Τέλο, ε, προτείνω να αυξηθεί λίγο το ποσό στη Διεθνή Συνεργασία για τη Φορολογία. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό, αν δει κανείς και τη συμφωνία στο G20. Τέλος, προτείνω να ξεκινήσει μια νέα προπαρασκευαστική ενέργεια για αύξηση ε, της δημιουργίας υποδομών ε, και της δημιουργίας ικανοτήτων των τελικών χρηστών και άλλων εμπλεκομένων φορέων για τις σημαντικονομικές υπηρεσίες σε συνέχεια το πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτή θα είναι μια πολύ μετριοπαθή συνεισφορά εκ μέρους μας για να αντιπαραταθούμε στο, στην άσκηση πιέσεων που γίνεται στον τομέα των μεταψωτικών υπηρεσιών. Σε ευχαριστούμε. Ο Σβέν τώρα εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστούμε μάλλον Σβέν. Θα δώσω λόγο στον κύριο Σφάμπ εκ μέρους του ΕΛΚ που αντικαθιστά το σκέφτεσαι γιατί. Mm. Όχι. Παρακαλώ. Δεν ήθελα να μιλήσω για το συνολικό πακέτο, αλλά να αναφερθώ στην τελευταία παρατήρηση του συναδέλφου Γκίγκολτ για τον προϋπολογισμό που είπε ότι πρέπει να τον αυξήσουμε ε, σε ε, ε, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ανεξάρτητους. Δεν είναι δυνατόν. 900.000 ευρώ έχουν πάρει από δημόσια κονδύλια αυτές δεν είναι δυνατόν, ε, δυσχεραίνεται έτσι η δουλειά μας ε, μέσα από finance swaps. Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι πρέπει να Οκ. Okay, uh, Mrs. McCarthy wants uh, the floor on this point. Um, well, um, I sincerely hope, colleagues, that you don't vote. Ελπίζω να μην ε, ψηφιστεί η σύσταση του κυρίου Λάγκεν εδώ, γιατί ως μέλος του Finance Watch ε, πρέπει να πω ότι αυτό δημιουργήθηκε ως οργανισμός για να επιτρέψει στους καταναλωτές και τους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για χρηματοδότηση, να καταλάβουν τον κόσμο της, το, της χρηματοδότησης και ε, εδώ έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά ε, για το λόμπινγκ από τις επιχειρήσεις ε, ύψους 10 ε, δις. Γιατί λοιπόν για οικονομικά θέματα να μην δώσουμε χρήματα για να ενημερωθούν οι πολίτες μας. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Λάγεν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χουάν Νιόκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ συμμερίζομαι σχεδόν το σύνολο των ε, απόψεων του κυρίου Γκίγκολτ. Οι τροπολογίες που υπέβαλα καλύπτονται τις συμβαστικές τροπολογίες του κυρίου Γκίγκολτ. Οπότε πραγματικά θέλω να επενέσω τη δουλειά που έγινε και όσον αφορά την τροπολογία 7505 θα συμφωνήσω μετά όσα είπε ο κ. Μακάρθη και η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων σήμερα δεν μπορεί να Ε, πάρει εμπειρογνωμοσύνη από οποιαδήποτε ομάδα πιέση για όλα τα θέματα συνολικά. Και εδώ πραγματικά είναι σημαντικό για τη μελέτη μα να έχουμε τέτοιου είδους ε, στήριξη και από ομάδε όπω η Finance Watch για την οικονομική μα διοργάνωση. Ευχαριστούμε κύριε Νουάνι. Ο κύριο Ντόρβαλτ γιατί του φιλελεύθερο Δεν είναι εδώ. Υπάρχει κάποιο από την Άλντε που θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Οπότε, εκ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Καμάλ. Θα πάρετε τον λόγο. Όχι. Is there Κάποιος άλλος από την ΚΟΕ. Κύριος Κλούτε. Κύριος να θα κάνω μερικές παρατηρήσεις ε, για την ΚΟΕ. Καταρχήν στηρίζουμε την έκθεση του Σβέν Γκίγκολ, πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλή, είναι σύντομη βέβαια. αυτή αυτές είναι οι επίσημες προδιαγραφές, οπότε προσπαθήσαμε να την υποστηρίξουμε με τις τροπολογίες και να τη βελτιώσουμε λίγο σε κάποια σημεία, αλλά γενικά συμφωνούμε με την έκθεση και μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ καλή. Τώρα, δύο παρατηρήσεις που θέλω να υπογραμμίσω ε, καταρχήν η πρικοδότηση των εποπτικών αρχών που είναι πολύ σημαντικό πράγμα γιατί αυτά που αποφασίζουμε και θέλουμε να εφαρμόσουμε σε κανονιστικό επίπεδο χωρίς εποπτικές αρχές που θα λειτουργούν αποτελεσματικά δεν γίνονται οπότε πρέπει να έχουν κονδύλια στη διάθεσή τους για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Το για το Finance Watch πρέπει να πω ότι στην αρχή αυτής της θητείας του Κοινοβουλίου από κοινού ε, συμφωνήσαμε ως Επιτροπή να δημιουργηθεί, να συσταθεί αυτή, αυτό το όργανο. Ε, τότε είχαμε ανθρώπους ε, ε, ως συμβούλους ε, από το κύκλο των λόμπις και των επιχειρήσεων και δεν είχαμε άλλους ανεξάρτητους. Δεν υπήρχε δηλαδή η δυνατότητα η κοινωνία των πολιτών να παίξει το ρόλο της εδώ, ενώ τώρα μπορεί, γι' αυτό το στηρίξαμε. Ακόμα και αν δημιουργεί περισσότερη δουλειά, συμφωνώ με τον κύριο Λάγκεν, περιπλέκονται έτσι τα πράγματα. Αλλά αυτός είναι ο λόγος και το νόημα αυτό του του Finance Watch ούτως ώστε να έχουμε εναλλακτικέ πηγές και να μπορούμε να βλέπουμε όλη την κάθε προβληματική μέσα από διαφορετικά οπτικά πρίσματα. Γι' αυτό συμφωνώ και εγώ και θα ήθελα να συμφωνήσουμε με τη διατύπωση του Σβέν Γκίγκολ σχετικά με αυτό. Σβέν, ο κύριος το λόγο. Θα του δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο και θα σας παρακαλέσω να είστε όλοι σύντομοι διότι πραγματικά έχουμε καθυστερήσει. Και μετά θα πάρετε πάλι το λόγο. Ε, κύριε Γκίγκολτ. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομο. Απλώς θέλω να πω ότι στηρίζω αυτό που είπε ο Σβέν Γκίγκολτ. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά διότι όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, ιδίως όταν συζητάμε για το μύθι, νομίζω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 200 διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι. Δεν λένε όλοι τα ίδια, αλλά οι καταναλωτές, εάν υπάρχουν καταναλωτές ε, καθόλου στην προοπτική την οποία εξετάζουμε, δεν είναι τόσο πολλοί. Ακόμη λοιπόν και κάποιες φορές διαφωνούμε, ίσως αρκετά συχνά με κάποιες από τις ομάδες, ε, χρήσιμο είναι σε δημοκρατικό πολίτευμα να τα συζητάμε αυτά και εγώ είμαι συνηθισμένο σε τέτοια στη χώρα μου μπορούμε να δεχτούμε ακόμη και τα επικρατικά σχόλια. Σα ευχαριστούμε κύριε Σμιτ. Η, η κυρία Λούλινγκ. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ να είστε και εσεί σύντομοι. Μια γενική παρατήρηση θα κάνω μόνο. Ξέρετε ότι πρέπει να κάνουμε εξοικονομήσεις. Και λάβαμε και σειρά μέτρων που μας πλήττουν και μας εγώ είμαι κοσμήτορ και γνωρίζω τα προβλήματα γιατί θέλουμε να μειώσουμε κατά 30% τα ταξίδια κλπ. Και εδώ πετάμε τα λεφτά από το παράθυρο. Οι άνθρωποι αυτοί χρηματοδοτούνται ήδη. Τι, γιατί ε, ε, θα πρέπει να λέμε ότι βοηθούν τις πολίτες. Έχουν ε, κάτι τεράστιους μισθούς και τώρα πρέπει να τους χρηματοδοτήσουμε ακόμα περισσότερο. Τη γενική γραμμή που έχουμε στο Κοινοβούλιο για τις εξοικονομήσεις, ε, γιατί δεν ισχύει, γιατί πετάμε από την άλλη λεφτά από το παράθυρο. Είμαι τελείως κατά. Ευχαριστώ. Τέλος ο κύριος Γκίγκολ, το εισηγητής. Συνάδελφοι, κατά πρώτον ευχαριστώ για τις ενισφορές σας, τουλάχιστον στις γενικές γραμμές του αν θα στηρίξουμε ή όχι το, τις ευρωπαϊκές ε, οικονομικές αρχές όπως τις αποπτικές αρχές και τη Eurostat νομίζω ότι υπάρχει εδώ ευρεία συνένεση. Αυτό χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα διότι διαφορετικά όλη η νομοθετική μας προσπάθεια θα αποδειχθεί τί. Σας ευχαριστώ λοιπόν κατά πρώτον γι' αυτό. Τώρα σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που έγινε για τους αριθμούς του προπολογισμού να ότι η δημοσιονομική αυτή γραμμή δεν είναι συγκεκριμένα για την χρηματοδότηση του Finance Watch. Είναι ανοιχτή προκήρυξη για όλους τους οργανισμούς που δεν ε, χρηματοδοτούνται από τον ίδιο κλάδο. Σήμερα η πρώτη πρωτοβουλία που θα χρηματοδοτηθεί για δύο χρόνια χρησιμοποιείται από δύο διαφορετικού οργανισμούς και ένας από αυτούς είναι εκπρόσωπος των χρηστών των χρηματοπιστωτικών αγορών. Κάτι που Ε, θα εξαρτηθεί πολύ από το πώς θα διαμορφωθεί η δική μας νομοθετική προσπάθεια. Τώρα, για τη χρήση των κονδυλίων στις Βρυξέλλες και για να ε, εκπροσωπηθούν σωστά τα ιδιωτικά συμφέροντα στις χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίες, εδώ έχουμε περίπου 300.000 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 700 ε, επαγγελματίες του χώρου του λόμπινγκ που προσφέρουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι αυτοί που περιμένουν αυτά τα κονδύλια. Είναι πολύ λίγα λοιπόν, διότι είναι πολύ δυσκολότερο να συλλέγονται χρήματα από 400-500 εκατομμύρια πολίτες, από ότι να τα συλλέγουμε από αυτούς που μπορούν να δώσουν και κάποιο κέρδος ε, και να μας δώσουν και κάποιο όφελος επηρεάζοντας την νομοθεσία μας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές δυνάμεις που πρέπει να εξισορροπηθούν και θα πρέπει να γίνει και σε άλλους τομείς της καταναλωτικής προστασίας, προστασία μάλλον των καταναλωτών, τη περιβαλλοντική προστασία. Στι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Ευτυχώ υπήρξε αυτή η διακομματική πρωτοβουλία που δημιούργησε αυτόν τον προπολογισμό εδώ και δύο χρόνια και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί. Ε, να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σε αυτή τη διακομματική πρωτοβουλία ένα βαθμό α, πρώτη κατηγορία μεταξύ του τι συστήνει ως προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει το Κοινοβούλιο. Αυτό το A λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντικό. Και για να το πω εδώ, εδώ στα, σε ωραία γερμανικά, είναι σαν να πετάμε από το παράθυρο αυτήν την ε, ευκαιρία που μας δόθηκε. Είναι απλό το θέμα λοιπόν και αφορά μια κατάσταση που ισχύει στην πραγματικότητα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εγώ λοιπόν θα έλεγα να υπερψηφίσουμε την ε, δημοσιονομική γραμμή 6705. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκίγκολντ. Πολύ γρήγορα να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Α, θα το ψηφίσουμε σε λίγα λεπτά. Σε λίγα δευτερόλεπτα μάλλον αφού δούμε το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξη, της ανακοινώσεις για τους ενεξελίξει τριμερείς διαλόγους. Έχουμε εδώ δύο τριμερείς διαλόγους που θα ξανάρχισαν στις 10 Ιουλίου για να ε, εγκρίνουμε την τεχνική αποτίμηση και τα τεχνικά μέτρα καθώς και τις μακροπρόθεσμες εγγύησεις τα συμπεράσματα και οι συζητήσει που έγιναν αντικατοπτρίζουν σωστά τι δικέ μα διαπραγματεύσει, όμω, χωρί εντολή του Συμβουλίου δεν μπορέσε να επιτελεστεί πραγματική πρόοδο. Επίση, έγιναν συζητήσει για μια, ε, την ανάγκη μια σύντομη και αποτελεσματική νέα οδηγία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το κενό που θα δημιουργηθεί από την 1η Ιανουαρίου τη ερχόμενη Χρονιά. Προτάθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2016 να έχει προβλεφθεί ε, ημερομηνία θέση σε ισχύ για αποτελεσματικότερη υλοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τροποποιήσει βέβαια δύο οδηγίες ε, με αυτή τη ε, διαδικασία. Στους τρομερούς διαλόγους μας είπε το Συμβούλιο ότι αν ε, προτείνει οδηγία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβάλλοντας την ημερομηνία στο 2016 θα συμφωνούσε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αναμένεται τώρα να εγκρίνει πρόταση πριν το τέλος του μήνα. Στον επόμενο, τους επόμενους τριμερείς διαλόγους θα τους έχουμε στις 10 Σεπτεμβρίου και 10 Οκτωβρίου. Σε ό,τι φορά το MIFID, δεύτερος τριμερείς διάλογος έλαβε χώρα χθες, όπου συζητήθηκαν ε, τα εμπορικά αγαθά και οι εξαιρέσεις. Ο επόμενος τομές διάλογος θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου. Για την οδηγία των ανακτήσεων έγιναν δύο γύροι ε, στις 10 Ιουλίου και στις 4 Σεπτεμβρίου. Συζητήθηκε αρχικά το πεδίο της οδηγίας και πώς θα πρέπει να εργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ στη δεύτερη συζήτηση συζητήθηκαν συμβαστικές προτάσεις για το πεδίο και ζητήματα για τις αρχές εξυγίανσης. Θα πρέπει να συνεχιστεί η τεχνική δουλειά σχετικά με το θέμα αυτό ενώπιση των επόμενων τριμερών διαλόγων. Ω προ τι συζητήσει μα με το Συμβούλιο για τι προτινόμενε εγγυημένε καταθήσεις και το σχετικό πρόγραμμα, ο εισηγητή για το θέμα αυτό λέει ότι θα πρέπει να ξαναρχίσουν οι συζητήσει για το θέμα αυτό παράλληλα με τι διαπραγματεύσει για το BIRD. θα πρέπει να εγκριθούν όλα αυτά μέχρι την Ολομέλεια του ε, Νοεμβρίου. Το, η Δημοτευτική Ομάδα του Κοινοβουλίου συναντήθηκε με τους υπευθύνους του Συμβουλίου στην αρχή αυτής της εβδομάδας και αποφασίστηκε να ξεκινήσουν οι επίσημες πολιτικές συζητήσεις τον Οκτώβριο οι ομάδε και του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να είναι σε θέση να συζητήσουν ε, τα ευαίσθητα ζητήματα μεταξύ τους κατά πόσο για να δουν κατά πόσο υπάρχουν επικαλύψει μεταξύ των δικών του προτεραιοτήτων. Simon, the rapporteur, want to get the floor. Nein, äh, nur einen Satz. Ich bin sehr froh. Χαίρομαι διότι η αναδιάρθρωση και η εξυγίανση προχωράνε καλά και μας δίνουν και περιθώριο να κινηθούμε κι εμείς. Βλέπουμε περιθώρια και στο Συμβούλιο. Οπότε ελπίζουμε ότι μετά από δύο χρόνια στασιμότητας λόγω στάσης του Συμβουλίου θα μπορέσει τώρα ο φάκελος αυτός να προχωρήσει ούτω ώστε αν πάνε όλα καλά να πάει το θέμα στην Ολομέλεια προς ψήφιση τον επόμενο Φεβρουάριο. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος αναλαμβάνει τώρα για να διεξαγάγει την ψηφοφορία. Thank um, Σε ευχαριστώ, Πάμπλο. Να προσθέσω μία μικρή ανακοίνωση η οποία αφορά τον ενιαίο μηχανισμό SSM σε ό,τι αφορά το επίπεδο πρόσβασης που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πρακτικά της συνεδρίασης του Επαπτικού Συμβουλίου δεν, ε, δεν έχουμε ακόμη ε, κάτι στα χέρια μας, αλλά περιμένουμε και μετά θα συνεχίσουμε. Στο επόμενο Στρασβούργο θα ψηφίσουμε για αυτόν τον ε, νέο αποπτικό μηχανισμό. Ελπίζω πάντως να έχω τα, ε, όλα τα στοιχεία σήμερα μέχρι τις 5. Είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Το ΕΠΤΑ έχει αναβληθεί. Οπότε πάμε στο σχέδιο γνωμοδότησης του Sven Γκίγκολτ. Είστε έτοιμοι. Εγώ δεν έχω την κάρτα ψηφοφορία. Τέλο πάντων θα το σχεδιάσουμε αν χρειαστεί. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι δεν έχουν. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δυστυχώς είναι αμφίροπο. Πρέπει να ελέγξουμε. Και εγώ ψηφίζω νομίζω. Α, ναι, έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Δεν έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία. Δεν ναι. Τώρα ναι, ωραία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Αν και πιστεύω ότι εγκρίθηκε. Ένρεξη ψηφοφορίας. Αν ψήσατε όλοι. Άλλο ένα συν υπάρχει. Βλέπω ότι τώρα βάζετε τις κάρτες. Λοιπόν, άρα εγκρίνεται. Τροπολογία 9, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όχι, εντάξει, να ελέγξουμε. είμαστε όλοι. Πω. 20 προς 20. Άρα καταπίπτει, απορρίπτεται. Είχατε δίκιο. Πάμε στη συμβιβαστική Β υπέρ. Κατά. Ε, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Θέλατε να ελέγξουμε τη 12. Αλήθεια. Καλά. Ε, ας το κάνουμε. Ψήσατε όλοι. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 τώρα υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ να προσθέσουμε ένα μείον εδώ ψηφίσατε όλοι απορρίπτεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική C ή Γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε αν και νομίζω ότι απορρίφθηκε ελέγχουμε την τροπολογία ένα μείον να βάλετε παραπάνω. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 22 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Εντάξει, δεν σηκώσετε και πολύ τα χέρια. Μια ψήφος υπέρ να προσθεθεί πέρας εγκρίνεται. 23 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μα εγκρίθηκε. 22 εγκρίθηκε. Ναι, αυτό είπα, λέει πρόεδρος. Δεν κατάλαβα, Αρλίν, τι πρόβλημα έχει ακριβώ τέλο πάντων. 24 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ποιο θέλετε να ελέγξουμε. Το 24, εντάξει. Στις ψήφους κατά να προσθεθεί μια ακόμη. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική δέλτα D. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο τη έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένα σαν παραπάνω να μπει. Ψηφίσατε όλοι. Η ψηφοφορία λίγη. Εγκρίνεται. 23 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, 7 αποχές. Και τώρα τι έχουμε, τις ε, τροπολογίες ε, για τον προπολογισμό. Λοιπόν, 6700 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6701 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6702 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6703 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6704 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 6705 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξω το 6705 προσθέτουμε μία ψήφο στις ε, θετικές 23 προς 12 εγκρίνεται 6706 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 14 υπέρ κατά Να ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται βέβαια. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήταν μέσα στη συμβιβαστική, ήταν συμβαστική 2. 6711 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6712 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6713 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να σου ξαναδώσω, Παύλο, τώρα το, λόγο και την Προεδρία για την έκθεσή σου. Sorry. No, this is... Oh, yeah. We move on to the next item. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης, που είναι η εξέταση του σχεδίου γνωμοδότηση για την ποινική προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη μέσω ποινικού δικαίου. Πρόκειται για γνωμοδότηση λοιπόν προ την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, που είναι η καθήλυνα αρμόδια. Θα τα πω όμω στα ισπανικά, επειδή εγώ είμαι συγητής. για να με καταλάβετε. Λοιπόν, η βασική ιδέα αυτής της έκθεσης είναι ο εξυγχρονισμός, η ενίσχυση και η εναρμόνιση του συστήματος κυρώσεων κατά της παραχάραξης του ευρώ και άλλων νομισμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικαθιστά τον κανονισμό 1338 2001 και είναι μια πρωτοβουλία την οποία υποστηρίζω και ιδίω σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των κυρώσεων. Η περίοδο κρίση πρέπει να χρησιμεύσει για να ενισχύσουμε τον αγώνα που δίνουμε κατά τη ε, απάτης και θα πρέπει να έχουμε στοχευμένες κοινέ δράσεις με στόχο το, να πετύχουμε, ε, να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Το ευρώ έχει πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομική, χρηματοοικονομική και πολιτική ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. άρα πρέπει να το προστατεύσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη, ε, σε αυτά τα πολύ δύσκολα, στι δύσκολε συνθήκες που ζούμε, εμπιστοσύνη λοιπόν στο ευρώ, στο νέο νόμισμα. Και γι' αυτό θα πρέπει να το προφυλάξουμε από ε, το κίνδυνο παραχάραξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο στόχο ε, των ε, τροπολογιών που υποβάλλω ε, είναι γιατί θέλω να έχουν όλες οι χώρες μέλη ε, τους ίδιους και τις ίδιες συνθήκες. Επίσης θέλω να ε, τονίσω ότι στόχος είναι να έχουμε μια συνεπή γραμμή με άλλες εκθέσεις της ΕΚΟΝ που έφυγαν τα ίδια ζητήματα. Επίσης, προσπάθησα να συμπεριλάβω την ιδέα ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δρουν από κοινού. Συγκεκριμένα, συγκεκριμένα οι τροπολογίες μου ε, είναι πρώτον να δημοσιοποιούνται οι κυρώσεις ώστε να είναι αποτρεπτικές οι ποινές και αποτελεσματικές βέβαια. Άλλες τροπολογίες έχουν ως στόχο την αναλογικότητα των ποινών να περιληφθεί αυτή η αρχή σύμφωνα και με τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας Υπάρχουν επίσης άλλες τροπολογίες ε, με στόχο να έχουμε ένα ευρύ ε, πεδίο εφαρμογής. Δηλαδή να περιλαμβάνεται παραχάραξη ε, των τραπεζογραμματίων και των νομισμάτων. Να μην εστιάζουμε όμως μόνο στο ευρώ αλλά και σε άλλα νομίσματα. και σε ό,τι αφορά ε, τις αξιόπινες πράξεις σε σχέση με μέσα και πρώτες ύλες παραγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων έχω καταθέσει τροπολογίες γεννής και της σχετικής νομοθεσίας και τέλος θα πρέπει να διαβιβάζονται ε, τα ε, στοιχεία των υπόπτων ως ε, προϊόντων παραχάραξης ή κυβδηλίας τραπεζογραμματίων και κερμάτων στα εθνικά κέντρα ανάλυσης κατά τη διάρκεια ένδικων διαδικασιών. Ας ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις, δεν ξέρω. Α, η κυρία Φερέρα δεν είναι εδώ, υπάρχει κάποιος. Υπάρχει ο κύριος Παδάρ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Yes. Ε, Apologizes from... Ε, Συγγνώμη ε, για λογαριασμό της Ελίζα Φερέιρα που είχε άλλες υποχρεώσεις. Εγώ θα μιλήσω εξ ονόματός της. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την δουλειά του αυτή στο σχέδιο γνωμοδότησης και συμφωνώ με τη γνωμοδότησή του. Η πρόταση της Κομισιόν είναι ευπρόσδεκτη. Η παραχάραξη νομισμάτων του ευρώ συγκεκριμένα ε, δημιουργεί πρόβλημα εμπιστοσύνης στα νομίσματα. Οι κυρώσεις διασφαλίζουν ότι αντιμετωπίζεται το θέμα εμπιστοσύνης. Η εναρμόνιση επίσης είναι ευπρόσδεκτη εδώ. Τώρα στα 28 κράτη-μέλη θα έχουμε ε, ποινικοποίηση της παραχάραξης ε, με φυλάκιση και θα προβλέπονται και ε, δυνατότητες και εργαλεία στους, στις ανακριτικές αρχές. Η, βελτιώνεται η πρόταση της Κομισιόν αναφέροντας την κοινοποίηση των καταδικών και ποινικοποιώντα την παραχάραξη ε, και κυβδηλία του ευρώ και άλλων νομισμάτων. Συμφωνώ λοιπόν με την Κομισιόν και με τις προτάσεις. Δεν πρόκειται να καταθέσω σημαντικές τροπολογίες στην γνωμοδότηση του εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πάνταρ. Για την Λίμπε η κυρία Γουλάρ. Ευχαριστώ. Σε αυτή τη φάση θα δω κι εγώ με περισσότερη λεπτομέρεια τις προτάσεις. Έχω την ε, εντύπωση ότι πάνε στη σωστή κατεύθυνση τοπολογίε. Όμω αισθάνομαι ότι κάπω έχουμε χάσει από τον ορίζοντά μα τον ε, με ύψιστο στόχο μα. Πάμπλο. Νομίζω ότι ετοιμάζουμε ένα πολύ κείμενο για την ε, ποινική προστασία του ευρώ. Όμως, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παραχάραξη, θα πρέπει να καταργήσουμε τα χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ. Αυτά είναι που παροτρύνουν το οργανωμένο έγκλημα να προχωρήσει η παραχάραξη. Είτε παραχαράσουν είτε όχι. Και ανοίγοντα ε, τα ντουλάπια του δικτάτορα Μπεναλή, είδαμε ότι είχε μεγάλα χαρτονομίσματα και παχυλά ποσά σε χαρτονομίσματα ευρώ. Λοιπόν, αυτό το κείμενο το αν είναι ή όχι η καλύτερη νομοθετική πρόταση θα το δω. Αλλά μήπως κάτι έπρεπε να κάνουμε για να αποφύγουμε και την ε, παραχάραξη σημαντικών τέτοιων ε, υψηλών ποσών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Αγκουλάρ. Εκμένως των Πρασίνων. Ο κύριος είναι ο ασχετής, δεν είναι εδώ. Ο κύριος Λάμπερτ. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω αγγλικά ή γαλλικά. Τι προτιμάτε. Και τα δύο καλά είναι, λοιπόν, θα μιλήσω γαλλικά γιατί αρκετά δικαιολογικό με τα αγγλικά σήμερα. Και ο πρόεδρος, ε, όπως είπε, θα έπρεπε να ακούσουμε τον κύριο Ταβάρε, αλλά θα τον αντιτεστήσω εγώ. Να σα πω λοιπόν ότι δεν έχουμε την πρόθεση να υποβάλουμε τροπολογίε, διότι μα αρέσει αρκετά η έκθεση όσο έχει, αλλά θα συμφωνήσω απολύτω με αυτό που είπε η Σιλβή για την παραχάραξη των χαρτονομισμάτων μεγάλων ποσών. Α ε, σκεφτούμε λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που τα χρειάζονται αυτά τα χαρτονομίσματα. Εγώ δεν έχω πιάσει ποτέ τέτοιο χαρτονόμισμα στα χέρια μου. Αλλά φαντάζομαι ότι άλλοι τα χρειάζονται. Και δεν νομίζω ότι είναι τα πλέον ε, κατάλληλα άτομα. Δεν έχω τίποτα άλλο να δηλώσω. Ευχαριστούμε κύριε Λάμπερτ. Εκ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστέ, σκιώδη συζητητή, ο κύριο Φόξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η εναρμόνιση όπω την προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και την ερμηνεία ε, ποινικών υποθέσεων με τον σωστό τρόπο και τον ίδιο τρόπο μεταξύ των κρατών που χρησιμοποιούν όλα το ευρώ. Παρ' όλα αυτά, δεν στηρίζω τι λεπτομέρειε για τι ελάχιστε ποινέ για ποινικά δικήματα, όπω τα ορίζει το άρθρο 5 τη οδηγία, διότι θεωρώ ότι εδώ υπάρχει υπερβολική παρέμβαση στην ε, εθνική κυριαρχία των καταμελών. Επίση, με απασχολεί το άρθρο 11. Είμαι πεπισμένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει στα κράτη-μέλη την πρόσβαση σε συνθήκη, την προσχώρηση μάλλον σε συνθήκη, ή το κατά πόσον θα αποφασίσουν για μια συνθήκη ή όχι. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσω επί, επί περαιτέρω με του συναδέλφου μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φόξ. Κάποιο άλλο θέλει το λόγο εισηγητής θα απαντήσω στα ισπανικά. Ε, λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους ε, για τις παρεμβάσεις σας. Να είστε βέβαια ότι θα τις λάβω υπόψη ναι. και βέβαια θα συνεργαστώ με όλους μαζί σας, με όλους ε, εσάς. Ιδίω λαμβάνοντα υπόψη τι προτάσει τροπολέγηση να τι λάβω για να τι συζητήσουμε. Θα ήθελα να σχολιάσω όμω κάτι που ανέφερε η κυρία Γκουλάρ σε σχέση με τα χαρτονομίσματα των 200 και 500 ευρώ. Σέβομαι και είναι θεμητή η ανησυχία σας. Νομίζω όμως ότι το πρόβλημα των ε, χαρτονομισμάτων των 200 και 500 ευρώ δεν είναι πρόβλημα παραχάραξης, αλλά ξεπλήματος χρήματος. Και εμείς ε, Ουσιαστικά εδώ στην έκθεσή μας περιοριζόμαστε στα θέματα της παραχάραξης του ευρώ και άλλων νομισμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιμένω ναι λοιπόν μένω ότι είναι θεμητή ανησυχία σας κυρία Γκουλάρ για το θέμα αυτό απλά έχω τις αμφιβολίες μου για το κατά πόσον είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στη συγκεκριμένη έκθεση που επαναλαμβάνω έχει να κάνει με θέματα παραχάραξης και όχι με θέματα ξεπλήματος χρήματος. Παρ' αυτά με τα χαράς να το συζητήσω διμερό μαζί σας, αλλά να συζητήσω και με τον κύριο Λάμπερτ που έδειξε ε, και αυτός ε, ότι ανησυχεί για το ίδιο θέμα. Είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Σε ό,τι αφορά την, την προθεσμία κατάθεσης είναι ε, τροπολογιών είναι η 10η Σεπτεμβρίου, 24 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσει η Επιτροπή Οικονομικών την έκθεση. Η ΔΕ Επιτροπή που είναι καθήλυνα αρμόδια, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ψηφίζει στις 3 Οκτωβρίου. Όσο για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη κάποια ημερομηνία. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 10, που είναι η εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για τη χορήγηση εγγύησης Ευρωπαϊκής στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης. Η συγκητής είναι ο κύριος Μάρτιν. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Μπόλς διότι το όνομα μπροστά σας παραμένει αυτό της κυρίας Μπόλς. Δεν μοιάζω όμως με την κυρία Μπόλς. Ο μόνος λόγος είναι η λοιπόν. Όχι, όχι, αστειευόμουν. Πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή τη σύντομη γνωμοδότηση σε αυτή τη φάση. Πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γραμματεία για όλη τη βοήθεια και ιδιαίτερος τη δική μου το, δικά, το δικό μου βοηθό, τον Γιωάννη Σαπ, ο οποίο πραγματικά μέσω των χρονικών περιορισμών και επειδή ε, ήταν πολύ ευρύ το θέμα που πρέπει να καλύψουμε, έχει γίνει εξαιρετική δουλειά πρέπει να πω. Ελπίζω και άλλοι συνάδελφοι ότι θα εκτιμήσουν αυτή την έκθεση. Θα μιλήσω γερμανικά τώρα αν δεν σα πειράζει. Περί πρόκειται λοιπόν πιθανές απώλειες της ε, Τράπεζας Επενδύσεων που χρηματοδοτεί επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε και προηγούμενη έκθεση για το πλαίσιο εγγυήσεων της ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Σημαντικά για μας σημεία σε αυτή τη γνωμοδότηση αναφέρονται αφενός στον κίνδυνο κερδοσκοπίας. Αυτό υπάρχει στην τροπολογία μου υπαριθμών 7. Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Τράπεζα Επενδύσεων να, στηρίζει με δικό της ρίσκο της ε, και να χρησιμοποιεί και τα εργαλεία της κεφαλαία αγοράς. Εδώ θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξουν άσκοποι κίνδυνοι και να ανοίξει πόρτα σε κερδοσκοπία. Ε, μετά για τα πρότυπα αναφοράς θα πρέπει πιστεύω και ελπίζω να συμφωνήσει η Επιτροπή μαζί μου η Τράπεζα Επενδύσεων συγκεκριμένα να υποβάλει αναφορές σχετικά με... Ε, τη συμμετοχή και τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Και πρέπει να υπάρχει και ένας κατάλογος που να δείχνει ποιος σε τελευταία ανάλυση θα είναι ωφελημένος από αυτές τις πιστώσεις. Οι 8 και 9 τροπολογίες αναφέρονται με τα, στα ενδιάμεσα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στην αρχή του έτους διαβάσαμε σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται η Τράπεζα Επενδύσεων ε, πολύ υψηλέ ε, αμοιβέ για τη διαμεσολάβηση. Δεν επιτρέπεται αυτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια θα πηγαίνουν στα προγράμματα τα ίδια και όχι σε υπέρμετρε χρεώσει που θα εξαντλούν τα κονδύλια και δεν θα πηγαίνουν εκεί που θέλουμε. Το επόμενο θέμα είναι το κλίμα, όπου η Κομισιόν η ίδια προβλέπει ότι τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού θα πηγαίνει για την προσαρμογή στο κλίμα και την προστασία του κλίματος. Αυτό είναι πολύ καλό και το υποστηρίζουμε. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να υπάρχουν όμως συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με το τι σημαίνει φιλικό προς το κλίμα, ε, η όλοι οι Αυστριακοί νομίζω είμαστε πεπισμένοι, είμαι πεπισμένος ότι δεν πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση πυρηνικών εγκαταστάσεων και εργοστασίων. δεν θα πρέπει δηλαδή να βοηθάει η Τράπεζα Επενδύσεων και να δίνει λεφτά για να παρατείνουν τη δραστηριότητά τους και λειτουργία τους αυτά τα εργοστάσια. Επίσης, οι απαιτήσει των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εδώ πιστεύω πρέπει να είναι βέβαιο ότι οι επενδύσεις της τράπεζας δεν θα οδηγούν σε μεταφορά θέσεων εργασίας εκτός Ευρώπης. Μην δίνει λεφτά για να ε, φεύγουν οι θέσεις εργασίας λόγω μετεγκατάστασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για το ΕΛΚ, ο Σκιώδης, κύριο Στολόγιαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την εργασία που έκανε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Εμείς στηρίζουμε την έκθεση. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεχίσει αυτή τη δραστηριότητα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ε, ε, η αξιολόγηση τριπλού αλφα της Τράπεζας Επενδύσεων, ούτως ώστε τα δάνεια αυτά προς τις τρίτες χώρες να είναι ε, όσο γίνεται με χαμηλότερο επιτόκιο Τώρα, εις ό,τι αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης, θα υποστηρίξω με τις περισσότερες τροπολογίες. Όμως, ε, έχουμε ένα θέμα να συζητήσουμε ακόμα στην πολιτική μου ομάδα και αυτό αφορά την τροπολογία 3, υπαριθμών 3, που αφορά το ότι δεν πρέπει να χρηματοδοτείται η πυρηνική ενέργεια ανάντι και κατάντι διαδικασίες και αποθήκευση πυρηνικών καυσίμων. Ε, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε στην ομάδα μου για να ε, καταλήξουμε κάπου. Υπάρχει και μια άλλη τροπολογία. Η τέσσερα η χρηματοδότηση από την Τράπεζα Επενδύσεων δεν πρέπει να συμβάλλει στην ε, μετεγκατάσταση θέσεων εργασίας εκτός Ένωσης. Βέβαια, δεν θέλουμε να φεύγουν θέσεις εργασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ξέρω πώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να συμπεριλάβει το στόχο αυτό στην πολιτική της. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που δεν είναι στην γνωμοδότηση, αλλά στο παράρτημα 3 νομίζω, με τον κατάλογο χωρών ε, δικαιούχων για τέτοιες εγγύσεις και εδώ υπάρχει και η Αρμενία. Λαμβάνοντας υπόψη τι τύχη είχε η απόφαση που ελήφθη σε επίπεδο κράτους της Αρμενίας σχετικά με την εμπορική ένωση με τη Ρωσία ε, και το Καζαχστάν που απορρίπτει ουσιαστικά την, ε, συμφωνία, την υπογραφή της συμφωνίας με την Ένωση, υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να δούμε αν θα παραμείνει στον κατάλογο αυτών η Αρμενία. Ευχαριστώ και για τους σοσιαλιστές. δεν υπάρχει κανείς, για τους φιλελεύθερους δεν υπάρχει κανείς, για τους πράσινους θα μιλήσει ο κύριος Λάμπερς. Ε, πώς το καταλάβατε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Χάνς Πέτερ Μάρτιν. Όλες τις τροπολογίες θα τις υποστηρίξουμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα βελτιώσουμε κάποιες από αυτές. Πρώτον, τι προγράμματα χρηματοδοτεί η Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό αφορά και την εξωτερική και την εσωτερική εντολή της. Ε, να είμαστε ξεκάθαροι, όταν πρόκειται για καινοτόμα προγράμματα ενεργειακά, οι άλλες τράπεζες λένε «Α, δεν ξέρουμε, είναι σύνθετα τα θέματα, δεν ξέρουμε τι ρίσκο συνεπάγεται, είναι πολύ επικίνδυνο». Οπότε οι τραπεζίτες λένε «Μπορούμε να ε, διαχειριστούμε τον κίνδυνο που γνωρίζουμε». Είναι συντηρητικές συνήθως οι τράπεζες. Ακούω και άλλες τράπεζες να λένε όταν ας πούμε αιωλικό πάρκο, α πούμε στην ανοιχτή θάλασσα ε, συζητείται, λένε δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε το επίπεδο κινδύνου, δεν μπορούμε να το αναλάβουμε. Ενώ μπορούν να πάνε ας πούμε για σταθμούς παραγωγής ενέργειας με άνθρακα ή και πυρηνικά, πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας ή μπορούν να πούν ότι α, δεν το κάνουμε αυτό αν δεν έχουμε κρατικές ενισχύσεις που είναι περίεργο ε, για τις... Ε, ε, ε, κρατικές επιχειρήσεις, αλλά πάντως οι συνήθεις τράπεζες χρηματοδοτούν τεχνολογία του 19ου και του 20ου αιώνα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ε, τράπεζα επενδύσεων για να κάνει τα συνηθισμένα. Υπ' αυτή την έννοια αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε ένα σχέδιο για σταδιακή πάυση, όχι να πούμε θα μειώσουμε μόνο όλη τη χρηματοδότηση στον τομέα της ενέργειας, και θα αυξήσουμε τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας, θα πούμε ότι ό,τι είναι παλιό δεν θα απασχολεί πια την Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί αυτή λειτουργεί με χρήματα του δημοσίου που πρέπει να είναι καταλήτης για αλλαγή και όχι ε, μια συνηθισμένη διαδικασία. Θέλουμε λοιπόν ένα σχέδιο για σταδιακή εξάλληψη ε, μη ανανεώσιμων ε, προγραμμάτων και επιδοτήσεων και θέλουμε η Τράπεζα Επενδύσεων σταδιακά να επικεντρωθεί μόνο στην μετάβαση, την ενεργειακή μετάβαση, την αλλαγή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θέλουμε ε, να είμαστε συνεπείς προς το άρθρο 21 της συνθήκης, δηλαδή να είμαστε συνεπείς προς τους στόχους εξωτερικής πολιτικής και συμφωνώ εδώ με τον κύριο Στολόγεν, γιατί αν κάποια κράτη αποφασίσουν ότι θα είναι καλύτερα να μην έχουν ε, καλή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το κάνουν. Αλλά ε, προς Θεού, γιατί θα πρέπει τότε εμείς να χρηματοδοτούμε προγράμματα σε αυτά τα κράτη. Τέλος, και αυτό είναι παλιό μας αίτημα, πιστεύουμε ότι η Τράπεζα Ανασυγκρότηση και η Ανάπτυξη δεν πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται. Υπάρχουν πολλά διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θα πρέπει να λάβει τη δουλειά την τωρινή η Τράπεζα Επενδύσεων και η Παγκόσμια Τράπεζα. Καλύτερα θα είναι έτσι και είναι περίεργο ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν διατηρούν ιδρύματα που δεν έχουν προστιθέμενη αξία όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. σύμφωνο απόλυτα μαζί σας, εκτός μικροφώνου και πραγματικά εδώ είμαστε, ταυτίζονται οι απόψεις μας. Πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι, πρέπει, ε, επειδή είμαστε επιφορτισμένοι να δαπανούμε τα χρήματα των φορολογουμένων, πρέπει να ε, εξορθολογικεύουμε ε, τις δαπάνες ε, ακόμα υπάρχει και εδώ στο Κοινοβούλιο σπατάλη χρημάτων. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τις δαπάνες μας ε, εμείς. Χαίρομαι που μου δώσατε ευκαιρία να το πω αυτό. Μόνο έτσι μπορούμε να, δώσουμε, να ζητήσουμε σε άλλους τομείς αύξηση της χρηματοδότησης. Πρέπει να τα λέμε και τα δύο. Και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λάμπερτ. Εκ μέρους της ECR το λόγο έχει ο κύριος Φόξ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Ιβο ε, Στρέιτσεκ δεν μπορεί να είναι εδώ. Θα με συγχωρήσετε όμως ε, Πρέπει να διαβάσω αυτό που γράφει και όταν λέω εγώ ε, εννοώ αυτός. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Μάρτιν για τη δουλειά του πάνω σε αυτό το έργο. Καλωσορίζω τις προτάσεις ε, τη Κομισιόν γιατί στόχος είναι να είναι καλύτερε δυνατότητες ε, χρηματοδότηση εδώ εκτός Ένωσης μέσω της ΕΤΕΠ και κυρίω χώρες τη Ανατολική και Νότιας Τερικής σχέση Εγώ στηρίζω τις περισσότερε τροπολογίες του εισηγητού και όπως και ο κύριος Στόλογιαν ανησυχώ για τις τροπολογίε 3 και 4. Σε ό,τι αφορά άλλα σημεία θα καταθέσω δικέ μου τροπολογίε με τις εξή αρχές βασικά. Πρώτα απ' όλα στηρίζουμε ε, τις ε, δραστηριότητες ε, της ΕΤΕΠ εκτός και εντός Ένωσης. Θα πρέπει να παρέχει κεφάλαιο στις ΜΜΕ. Θα πρέπει επίσης τακτά να αξιολογεί το κόστος και όφελος ε, ε, των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για να δει την οικονομική τους βιωσιμότητα και το κατά πόσον συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως και σε προηγούμενα αιτήματα της ΕΚΟΝ ε, θα πρέπει στην ιστοσελίδα της εφόσον χρειάζεται να παρέχει τις πληροφορίες για τους διατόχους τους στα μακροπρόθεσμα δάνεια και να τηρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και να βλέπουμε τι κεφάλαια έχουν δοθεί, σε ποια περιοχή και για ποιο τομέα της βιομηχανίας. Τέλος, θεωρούμε ότι θα πρέπει η χρηματοδότηση της ΕΤΕΠ να έχει ως στόχο και την προώθηση ενός αποτελεσματικού ενεργειακού μείγματο. Να έχουμε διαφοροποιημένες δηλαδή πηγές ενέργειας στην Ένωση και έναν ασφαλή ενεργειακό, ε, μια ασφαλή αλυσίδα ενεργειακού εφοδιασμού. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φόξ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Άρα θα δώσω το λόγο για μία ακόμη φορά στον εισηγητή κύριο Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λάμπερτ που μόλις ε, ε, φεύγει για την προοδευτική του τοποθέτηση και την προοδευτική του προσέγγιση. Θα προσπαθήσω να συνδυάσω τη δική σας ε, θέση με των ε, υπολείπων. Ε, σίγουρα με την πυρηνική ενέργεια θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Θέλω να σας επενθυμίσω όμως ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη αυτό που είπε ο κύριος Λάμπερτ, ότι δηλαδή εάν δεν αποτελεί για μας κοινό στρατηγικό στόχο να δούμε προς το μέλλον και όχι μόνο να ε, δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, πρέπει δηλαδή να ε, εγκαταλείψουν σταδιακά κάποια τα κτλ. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες σας θα τις μελετήσω. Οι σοσιαλιστές δεν έχουν ακόμη ε, κοινοποιήσει την άποψή τους και επειδή έχουμε κάνει επιτυχημένες ε, συναντήσεις κατά το παρελθόν θα συγκαλέσω μία ακόμη για να μπορέσουμε να συστήσουμε και να καταλήξουμε στις συμβαστικές προτάσεις. Πρώτος, ευχαριστούμε κύριε Μάρτιν. Προθεσμία κατάρτιση τροπολογιών 19 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου. Οπότε και θα ψηφίσουμε. Τώρα, ε, η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου, ενώ δεν ξέρουμε πότε θα ε, ψηφιστεί έκθεση στην Ολομέλεια. Επόμενε μέσα διάταξης. Διάφορα. Δεν υπάρχουν διάφορα. Άρα εδώ μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Θα σας πενθυμίσω απλά ότι η επόμενη θα λάβει χώρα στις 16 Σεπτεμβρίου από τις 3 η ώρα μέχρι τις 6 και μισή το απόγευμα και την 3η 17 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 και μισή το μεσημέρι και από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6.30. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.